Colleagues, Συνάδελφοι, κύριε Μποστινάρου, ας ξεκινήσουμε σας παρακαλώ τη συνεδρίαση. Σα παρακαλώ, α αρχίσουμε τη συνεδρίασή μα Πρώτο σημείο τη σημερινή συζήτηση είναι οι ανακοινώσει τη Πρόεδρου σχετικά με τι αποφάσει των συντονιστών που συνεδρίασαν σήμερα το πρωί. Οι συντονιστές ε, όσον αφορά την ανάθεση τη έκθεση για την αναθεώρηση για την οδηγία για την αξιολόγηση περιβαλλοντικού αντικτύπου αποφάσισαν να αναθέσουν την έκθεση στην ομάδα τη ΓΚΟΕ για τη συνέχεια που θα δοθεί στι εργασίε. Ε, όσον αφορά το αέριο σχιστόλιθο έχουμε αφήσει ανοιχτή τις αναφορές εν ώψη μιας νέας εξέτασης των αναφορών αυτών γιατί θα παρακολουθήσουμε τις εξελέξεις των δραστηριοτήτων της ε, ΕΝΒΙ και της ΙΤΡΕ. Τώρα όσον αφορά την ακρόαση και τη σύνοδο που θα γίνει στις 5 Δεκεμβρίου μετά από πρωτοβουλία του Φόρουμ ε, για τις ειδικέ ανάγκες ε, θα προβλέψουμε μια συμμετοχή όμως ακόμα αναμένουμε την επισημοποίηση του προγράμματος, την οριστικοποίηση του προγράμματος από πλευρά του Φόρουμ που ανέλαβε αποκλειστικά την πρωτοβουλία και μετά θα το συζητήσουμε με τους συναδέλφους και θα τους ανακοινώσουμε και τις λεπτομέρειες. Εν πάση περιπτώσει ε, ήταν μια πρόταση από πλευράς του εκπροσώπου της ΓΚΟΕ να εισαχθεί στην παρέμβαση από πλευράς της Επιτροπής Αναφορών και μια εκτίμηση του αντικτύπου της οικονομικής κρίσης όσον αφορά τους ανθρώπους που ε, πάσχουν από κάποια αναπηρία το θέμα της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας που είχε προβλεφθεί για τις 19 Φεβρουαρίου εξετάστηκε, αλλά οι εργασίες της οργάνωσης είναι ακόμα υπό εξέλιξη, οπότε μιλάμε ακόμα για ένα σχέδιο και καθώς θα προχωράμε με τον καθορισμό του προγράμματος θα ενημερώσουμε τους συναδέλφους. Για τα διάφορα έχουν ε, εισαχθεί από τους πράσινους η πρόταση για πρόσκληση του Επιτρόπου Αντιπροέδρου Σεύκοβιτς για μια ακρόαση για το θέμα της ε, σωστής διαχείρισης για να υπάρξει και μια ενημέρωση για την κατάσταση έγκρισης του νέου κανονισμού για την ορθή διαχείριση. Επίσης, ακόμη μια φορά αναβλήθηκε η συζήτηση για την υπόθεση μιας εσωτερικής νομοθεσίας για τον εσωτερικού κώδικα μάλλον για την Κομισιόν για τις ερευνητικές αποστολές. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα εξεταστεί στη διάρκεια της επόμενης συνόδου, πιθανότατα με βάση την πρόταση που υποβλήθηκε πριν από κάποιους μήνες από το ΕΛΚΑ. Τέλος, η ομάδα του ΕΛΚΑ ζήτησε να λάβει από την ε, Γραμματεία πληροφορίες σε σχέση με το 7ο Φόρουμ για τα δικαιώματα των παιδιών, φόρουμ που διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για το οποίο είχε προβλέπεται Ε, που θα λάβουν την πρόσκληση. Περιμένουμε λοιπόν ενημέρωση από τη γραμματεία. Δεν υπάρχουν άλλες ανακοινώσεις. Ε, θεωρώ πως εγκρίνεται τις, ε, τα συμπεράσματα των συντονιστών και θα περάσω στο επόμενο θέμα, το σημείο 13 που είναι οι αναφορές 1252 του 2011 που έχουν έχουν υποβληθεί από τον κύριο Γκαλάσο και ο ΣΝΑΤΟ και η 88 του 2012 που υποβλήθηκε από την κυρία Ντάρια Μπονφιέτη. Η πρώτη υπογράφεται από, συνοδεύεται από 96 υπογραφές και οι δύο αφορούν τα δικαστικά πορίσματα σε σχέση με την αεροπορική καταστροφή της Ούστικα. Ειδικά η δεύτερη αναφορά αναφέρεται στη δυσκολία που έχουν αντιμετωπίσει οι έρευνες για να φτάσουν στην αλήθεια ώστε να ξεκινήσουν εξεταστικές επιτροπές διεθνείς και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι παρούσα η κυρία Μπομφιέτη, στην οποία δίνω πέντε λεπτά. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, αξιότιμη κυρία Ευρωβουλευτέ, σας ευχαριστώ και όλους και την Πρόεδρο για την διάθεσή σας και για την προσοχή σας. Θα ήθελα καταρχήν να σας πω πώς δεν βρίσκομαι εδώ για να κατηγορήσω οποιονδήποτε, αλλά για να ζητήσω και να επιστήσω την προσοχή σας στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Ιταλική Εισαγγελία ώστε να ρίξει φως σε ένα δραματικό ατύχημα και για να το πω καλύτερα θυμίζοντας τα λόγια του ίδιου σας του Προέδρου, του Μάρτιν Σούλτς, έτσι ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμμετέχει στις ε, λυπηρές και περίπλοκες περιστάσεις ε, που αφορούν την καταστροφή της Ούστικα. Αυτό το λέω για προσωπικούς λόγους αλλά και λόγω της διαπίστωσης ότι αυτό το λυπηρό γεγονός δεν θα πρέπει να θεωρηθεί μόνο Ιταλική υπόθεση. Στις 19 και 27 στις 19 η ώρα φεύγει από, την Πολόνια για το Παλέρμο με 81 ανθρώπους, ε, με 81 επιβάτες, ένα αεροπλάνο το οποίο χωρίς κανένα λόγο εξαφανίζεται από τις οθόνες του ραντάρ και από τις πύργους ελέγχου ε, δυστυχώς το αεροσκάφος αυτό χάθηκε με, έπεσε με 81 θύματα. Για πολλά χρόνια ε, επικράτησε αβεβαιότητα λόγω της, ε, του ότι τα Ιταλικά πολεμικά αεροσκάφη υποστήριξαν στις επίσημες τους ανακοινώσεις ότι το αεροσκάφος έπεσε λόγω δικής του βλάβης ε, μέσα σε καθαρό ουρανό, ε, ενώ δεν υπήρχε δηλαδή κανένα εμπόριο. Εγώ μπόρεσα να ισχυριστώ και υπάρχουν ε, οι καταγραφές των ραντάρ. Δυστυχώς, τα πρώτα χρόνια της σιωπής Καταστράφηκαν πολλά στην Ιταλία και γι' αυτό θα ήθελα ακόμα και σήμερα να υπογραμμίσω τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας. Θέλω να θυμίσω ότι λόγω μιας συνεργασίας του ΝΑΤΟ, μιας ομάδας εμπειρογνωμόνων του ΝΑΤΟ με έναν Ιταλό δικαστή που είχε αναλάβει τη δική μας υπόθεση, αυτός ο ουρανός ο οποίος υποτίθεται ήταν τελείως καθαρός και χωρίς καμιά παρουσία αεροσκάφους ο ίδιος ο Ιταλός δικαστής τελικά το 1999 υποστηρίζει το εξής και παραθέτω το ατύχημα αυτό ε, συνέβη μετά από στρατιωτικές σχήσεις ε, αναχέτησης αυτό το αεροσκάφος ε, κατερρύφθη μέσω, με 81 θύματα. Ήταν ένα, μια, μια ε, ενέργεια πολεμική. Ήταν μια επιχείρηση συγκαλυμμένη κατά της ε, χώρας μας, ε, μια διεθνής δηλαδή συνωμοσία στην οποία καταρρίφθηκαν όρια, ε, σύνορα και δικαιώματα. Δεν δόθηκε καμιά εξήγηση για τα όσα έχουν δοθεί, έχουν συμβεί. Παραβιάστηκαν τα σύνορα και τα δικαιώματα, όχι μόνο της Ιταλίας, αλλά ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα θεωρώ αυτή την τραγωδία και ξανακολουθώ να το επαναλαμβάνω, όχι μόνο Ιταλική, γιατί Υπάρχουν ψεύδι, ψευδείς μαρτυρίες, καταστροφή αποδείξεων και εξακολουθούν να λείπουν οι απαντήσεις ή να είναι οι απαντήσεις ελλειπείς της Γαλλίας, της Γερμανίας και του Βελγίου. Το αεροσκάφος ε, είχε πορεία στα σύνορα της, ε, των, των Ιταλικών συνόρων που είναι όμως και σύνορα ευρωπαϊκά όπου κυκλοφορούν αεροσκάφη και πλοία κάθε εθνικότητας. Ε, πέρα από τα αεροσκάφη που το ίδιο το ΝΑΤΟ ακόμα και σήμερα δεν μπορεί να εντοπίσει πετούν αεροπλάνα αμερικανικά, λιβικά αλλά και ευρωπαϊκά, βελγικά και γερμανικά. Και θυμίζω ότι ο πρόεδρος Κωσίγκα μετά από υποδείξει των Ιταλικών μυστικών υπηρεσιών έριξε τις υποψίες στις γαλλικές μυστικέ υπηρεσίε τα τελευταία χρόνια της ζωής του και να θυμίσω ότι η Ευρώπη πάντοτε πιο σοβαρά ε, ε, αντιμετώπιζε αυτή την αντίθεση ανάμεσα στο βορρά και στο νότο, ενώ παρέμενε συγκαλυμμένος και ο πόλεμος, η, έχθρα ανάμεσα στο, στον ε, Ανατολή και στη Δύση. Στην ε, στην Περσία υπάρχουν αμερικανικές δυνάμεις, Ιράκ, Ιράν, παροχή πυρηνικών υλικών, διαρκώς ανησυχητικός ε, είναι ο ρόλος της Λιβύης, ε, αυξάνονται οι εντάσεις με το το μεταξύ υπάρχουν ε, συγκρούσεις και ανάμεσα στη Λιβύη και την Αίγυπτο και ο πρόεδρος Σαντάτ ορίζει καθεστώς επίγουσας ανάγκες ανάμεσα στις δύο χώρες και ζητά στήριξη αμερικανική για την Αίγυπτη. Θα ήθελα να λάβετε υπόψη ότι λόγω αυτών των διεθνών εντάσεων που ενδιαφέραν ιδιαίτερα την Ευρώπη και όχι μόνο την Ιταλία, πολλές στρατιωτικές πτήσεις που ήταν ένοπλες ε, και διέσχιζαν τα ουρανούς μας. Υπάρχουν ένα σωρό σενάρια τα οποία έχουν προταθεί, ότι δηλαδή καταδίωκαν κάποιο αεροσκάφος του Καντάφη ή και τα λοιπά. Και πρόκειται για υπόθεση ευρωπαϊκή, γιατί ακόμα και σε αυτό το, μέσα σε αυτό το διεθνές σκηνικό δεν μπορούμε να θεωρήσουμε πως είναι μόνο ιταλικά τα δικαιώματα στη ζωή, στη διάσωση και στην ασφάλεια των μεταφορών. Και εν τέλει και στην υπεράσπιση των συνόρων. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που μας παρουσιάσατε αυτή την αναφορά και θα δώσω το λόγο στον Τόμας Κοσούτο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ελπίζω ότι θα προσθέσει κάτι σε σχέση με το δικό μας σχόλιο ανικανότητας το οποίο <clears throat> έχουμε τεκμηριώσει και γραπτός. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Συγγνώμη, δεν μιλάω Ιταλικά και έτσι δεν μπορώ να απαντήσω στα Ιταλικά, θα σας μιλήσω αγγλικά. Θα ήθελα να υπενθυμίσω πως η Κομισιόν γνωρίζει την υπόθεση της Ουστίκα πάνω από 30 χρόνια μετά από το, από όταν συνέβη αυτή η τραγωδία γνωρίζουμε ότι και τα θύματα περιμένουν δικαιοσύνη Φοβάμαι όμως πως υπό τη συνθήκη της Λισαβόνας η κατάσταση παραμένει η ίδια. Η Κομισιόν δεν έχει αρμοδιότητα να παρέμβει στη λειτουργία των συστημάτων δικαιοσύνης ε, των κρατών μελών. Αυτό είναι αρμοδιότητα των αρχών των κρατών μελών. Η Κομισιόν λυπάται για το ότι η Κομισιόν και άλλα δύο κρατημέλη δεν έχουν ακόμα κυρώσει την σύμβαση 29 Μαΐου, 2000 για συνεργασία σε ποινικά θέματα που ήδη ισχύει σε 24 κρατημέλη. Θα ήθελα επίσης να υπενθυμίσω πως η Κομισιόν έχει παρουσιάσει ένα συνολικό πακέτο μέτρων για την ε, προστασία θυμάτων εγκλήματος. Υπάρχει οδηγία για τα δικαιώματα των θυμάτων ε, εγκληματικών ενεργειών που υιοθετήθηκε από Συμβούλιο και Κοινοβούλιο το φθινόπωρο αρχές Οκτωβρίου και θα ισχύσει σύντομα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ παρόλα αυτά. Υπάρχουν παρεμβάσεις από πολλές των συναδέλφων. Μπουστινάρο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε με μια περίπτωση η οποία είναι πραγματικά συγκλονιστική. Γιατί πρόκειται για κάτι το οποίο δεν υπάρχει α, αναλογό του στην ευρωπαϊκή ιστορία. Πρόκειται για θύματα, πολίτες, ενός ατυχήματος εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μιλάμε για το κομμουνιστικό μπλοκ, γιατί θα μπορούσε να έχει συμβεί και εκεί κάτι τέτοιο. Και, βεβαίω. έχουμε την συσκότηση των γεγονότων που οδήγησαν σε αυτή την τραγωδία. Κουκούλωμα, σιωπή, γύρω από αυτή την υπόθεση και βεβαίω έτσι ε, αμφισβητείται η αξιοπιστία οποιασδήποτε διαδικασίας. Δηλαδή, αποφάσεις παραδείγματο χάρη των ε, δικαστηρίων ή τυχόν προσφυγές για την περιουσία των αεροπλάνων. Αλλά εδώ πέρα μιλάμε για ένα πολιτικό αεροσκάφος το οποίο πέφτει από τον ουρανό για άγνωστους λόγους ή τεχνικούς λόγους όπως είπαν και κανείς δεν ξέρει τι έγινε. Σε εποχές που έχουμε δορυφόρους, ραντάρα και ελέγχεται ο εναέριος χώρος, ο θαλάσσιος χώρος, η γη έχει τεχνικά μέσα η Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν αντιλαμβανόμαστε γιατί δεν έχει γίνει τίποτα. Τουλάχιστον ένα φυσιολογικό πρόσωπο, ένας κανονικός άνθρωπος όπως εγώ. Και εδώ πέρα Βεβαίως αμφισβητείται η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν 30 χρόνια, δεν μπορούν, 30 χρόνια μετά δεν μπορούν να μάθουν οι συγγενείς τους γιατί πέθαναν αυτοί οι άνθρωποι. Ε, τεράστιο πρόβλημα. Δεν είναι μόνο θέμα πολιτικών αποφάσεων επιλογών. θα μπορούσαν να γίνουν ε, διάφορες ε, έρευνες ε, για να βρεθεί μια απάντηση. Θα ήταν δυνατόν, αλλά η απάντηση της Κομισιόν είναι απαράδεκτη. Γιατί, επαναλαμβάνω, μιλάμε για ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ο γεγονός πως ένας Ιταλός δικαστής Ε, αμφισβητεί έτσι την αξιοπιστία των θεσμικών οργάνων της ε, χώρας του με το να αρνείται να συνεργαστεί σε μια τέτοια περίπτωση και αυτό είναι μια είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να μας αφήσει ε, ασυγκίνητους Εντάξει, μπορεί να πει κανεί πω περάσαν 30 χρόνια, τι να ψάχνουμε τώρα. Δεν είναι σωστό αυτό. Εδώ πέρα έχει δίκιο. Δεν ήξερα αυτή τη δήλωση του Προέδρου του Μάρτιν Σούλτς, αλλά τη χαιρετίζω. Γιατί θεωρώ πως ε, πρέπει να ασκήσουμε πίεση στις Ιταλικές ε, αρχές για να ε, σηκωθεί αυτό το πέπλο μυστικότητας. Αλλιώς υπάρχει εντύπωση πως θέλουν κάποιοι να αποκρύψουν την αλήθεια, να μην μάθουμε τι συνθήκες που οδήγησαν σε αυτή την τραγωδία, να μην μάθει τίποτα το κοινό. υπάρχουν ε, πολιτικο-στρατιωτικές συνθήκες. Υπήρχαν και τότε. Και το αντιλαμβάνομαι αυτό σε έναν βαθμό. Υπήρχαν δηλώσεις ε, του τότε εκπροσώπου του ΝΑΤΟ ε, για τον πόλεμο της Ιουγκοσλαβίας που μίλησε για παράπλευρες απώλειες, αλλά πραγματικά το, το έτος 2012 είναι απαράδεκτο αυτό. Και πρέπει η Κομισιόν να καταβάλει κάποιες προσπάθειες και να κάνει τα θεσμικά εκείνα να κάνει τις σεισμικές κινήσεις ενέργειες έτσι ώστε οι Ιταλοί πολίτες να μάθουν τις αιτίε αυτής της τραγωδίας. Δεν μπορούμε τώρα πια να διαπιστώσουμε ποιος ήταν ο δράστης. Αλλά μπορούμε τουλάχιστον να απαιτήσουμε την τήρηση του νόμου. και οι άνθρωποι αυτοί, οι Ευρωπαίοι πολίτες, να έχουν δικαίωμα σε μια δίκαιη δίκη να μάθουν την αλήθεια. Δεν είναι δυνατόν να το κρύβουμε άλλο. Και η Κομισιόν ήταν πάρα πολύ προσεκτική ε, αυτό το καλοκαίρι, ειδικά όσον αφορά την παρακολούθηση της ε, πολιτικής κατάστασης στη Ρουμανία. Και δικαίως, αλλά θέλω να είναι εξίσου προσεκτική και με την περίπτωση αυτή και τον θάνατο αυτών των Ιταλών πολιτών. Η τραγωδία αυτή δεν επιτρέπεται να είναι μια σελίδα, μια υποσημείωση της, ε, της ιστορίας. Πρέπει να κινητοποιηθεί η Κομισιόν γιατί υπάρχουν μέσα τρόποι, αποδείξεις να βρούμε την ε, αλήθεια, υπάρχουν ε, διάφορα πρωτόκολλα, μια σειρά τεχνικών δεδομένων που μπορούμε να εξετάσουμε για να βρούμε μια κάποια απάντηση. Δεν μπορούμε νομίζω να έχω καμία... Δεν μπορούμε να έχουμε καμία άλλη θέση, θεωρώ. Και με συγχωρείτε να ακριβώς αλλά είναι πραγματικά τραγωδία. Γιατί μην ξεχνάμε πως και η Ευρώπη τότε ήταν χωρισμένη σε δύο μπλοκ, το ανατολικό και το δυτικό και ξέραμε πως υπήρχαν συγκρούσεις μεταξύ του ανατολικού και του δυτικού, αλλά εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης τότε ε, πέθαιναν Ευρωπαίοι πολίτες και δεν ήταν κανείς υπεύθυνος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Καρόνα. σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω αυτήν την Επιτροπή όλος ιδιαίτερος και εσάς κυρίως για την προσοχή που, δώσατε σε αυτή την υπόθεση που όπως θύμισε ο συνάδελφος Μποστινάρου είναι μια υπόθεση που, θα, που αξίζει μια απάντηση μετά από 30 χρόνια από την τραγωδία. Και οφείλω να πω και από αυτή την άποψη μέσα στα όρια των κινήσεων της κυβέρνησής μας και μέσα στα όρια μιας ε, τέτοιας ε, κατάστασης όπου ναι η Κομισιόν δεν έχει αρμοδιότητα διότι πρόκειται για θέματα εθνικά δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι και στη σημερινή απάντηση εντοπίζεται μια προφανής αδυναμία. Μια αδυναμία εξαιρετικά γραφειοκρατική απέναντι σε αυτή την υπόθεση. Θα περιμέναμε κάτι περισσότερο από πλευρά της Κομισιόν, γιατί ενώ το Κοινοβούλιο και μέσω αυτής της ε, ακρόασης της Επιτροπής Αναφορών έκανε κάποια εργασία πάνω σε αυτή την ε, υπόθεση, θα περιμέναμε από πλευρά τη Κομισιόν μια στάση λιγότερο γραφειοκρατική, θα έλεγα και κάπως πιο προσεκτική απέναντι σε μια υπόθεση που στην ουσία τι, τι ζητάει μια αυτή η αναφορά. Μετά από 30 χρόνια ζητάμε να δούμε τι ακριβώς συνέβη και για να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό είναι απαραίτητο οι χώρες Όντως, έχουν περάσει 30 χρόνια. Οι χώρες που έχουν πληροφορίες να τις δώσουν στη διάθεση της Ιταλικής Εισαγγελίας, ώστε να μπορέσουμε να δούμε επιτέλους τι συνέβη σε εκείνη τη τραγική μέρα και στιγμή. Εμείς θα συνεχίσουμε ως βουλευτές, αλλά Μπορούμε να ζητήσουμε και από την Κομισιόν να κάνει κάτι παραπάνω, εκτός από το ότι διαπιστώνει πως δεν έχει αρμοδιότητα. Και άρα να αναζητήσει τρόπους ε, για να ζητήσει από τα κράτη-μέλη να συνεργαστούν με την Ιταλική Εισαγγελία για να διαφωτιστεί επιτέλους υπόθεση. Και πάλι ευχαριστώ για την προσοχή που δίνει στο θέμα η Επιτροπή μας. Υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις. Όχι. Κανείς άλλος δεν ζητά το λόγο. Η αναφέρουσα της, της ε, αναφοράς τούτης έχει το δικαίωμα να απαντήσει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω όλους όσους θέλησαν να παρέμβουν. Συμφωνώ με τον κύριο Καρόνα. Πιστεύω ειλικρινά πως σε τούτη η Επιτροπή μπορεί να βρει άλλους τρόπους και άλλες μορφές για να παρέμβει. Μη ζητάμε με μια υπόθεση που πολύ γρήγορα προσπάθησα να σα εξηγήσω και που δεν είναι μόνο εθνική υπόθεση, να μας βοηθήσετε ώστε να δούμε ποιοι είναι επιτέλους υπεύθυνοι. Εμείς γνωρίζουμε και θέλω να επαναλάβω τι συνέβη. Οι εισαγγελείς μας κατάφεραν μετά από τόσα χρόνια και τόσες προσπάθειες και καταστροφές στοιχείων να καταλάβουν τι συνέβη εκείνο το βράδυ. Εκείνο το αεροσκάφος κατερρίφθη στα Ιταλικ, μέσα στο, Ιταλικό αεριοχώρο χώρο, στα σύνορα με το Διεθνή αεριοχώρο χώρο. Όμως είναι επίσης σαφές ότι δεν έφταιγε η Ιταλία. Ε, σε τι έφταιγε η Ιταλία, στο ότι εμπόδισε τους εισαγγελείς να δουλέψουν σωστά. Για πολλά χρόνια θα μπορούσα και να προχωρήσω και να μιλάω για ώρες για να σας διηγηθώ όλες τις ε, παραβιάσεις ε, τις οποίες προέβησαν τα θεσμικά όργανα της χώρας μου. Αλλά σήμερα ζητάμε τη συνεργασία έτσι ώστε οι δράστες που είναι διεθνείς και Ευρωπαίοι είναι ή η Γαλλία ή η Αμερική ή η Λιβύη ή το Βέλγιο ή η Γερμανία να, μπω, να μην πω ονομαστικά όλους τους υπευθύνου, αλλά η παρουσία εκείνων των αεροσκαφών, αυτών των διεθνών και ευρωπαϊκών αεροσκαφών είναι συμβεβαιωμένες πια, ε, βεβαιωμένη πια. Δεν χρειάζεται να το κουράζουμε πολύ. Το πράγμα είναι ευρωπαϊκό και διεθνές. Το λέει ο Ιταλός δικαστής και το γνωρίζουμε ήδη, δεν χρειάζεται να προσθέσουμε τίποτα άλλο. Ήταν ένα ε, συμβάν μιας ε, μάχης, αεροπορικής μάχης ε, στην οποία συμμετέχουν αεροσκάφη οπλισμένα με στρατιωτικές διαταγές. Αυτές, αυτά ήταν τα αεροσκάφη, τα στρατιωτικά αυτών των χωρών. Η παρουσία τους στον ουρανό είναι βεβαιωμένη πλέον. Απλώς θέλω να σας ζητήσω να βοηθήσετε ώστε οι χώρες αυτές του περιορισμού τη Ιταλία τι αναφέραμε, αυτέ οι χώρε να συνεργαστούν με την Ιταλική Εισαγγελία, όπω μόλι είπε και ο κύριο Γκαρόνα. Ευχαριστώ. Σα Σας ευχαριστώ και εγώ και ευχαριστώ του συνάδελφου που πήραν το λόγο. Σίγουρα δεν μπορώ να εκτιμήσω τη θέση της, ε, να χαρακτηρίσω και τη θέση της Κομισιόν ε, πολύ γραφειοκρατική. Το είπαν και οι συνάδελφοι που παρενέβησαν για αυτές τις λιγοστέ ε, φράσεις. Εξάλλου Είναι τελείως επιφανειακή αυτή η αναφορά, η οποία δεν στέκει κιόλα. Η αναφορά στο πακέτο μέτρων που στόχο έχουν να βοηθήσουν τα θύματα της, ε, του οργανωμένου εγκλήματος. Γιατί εδώ <laughs> δεν είμαστε εντός θέματος. Σίγουρα δεν μας ευχαριστεί το γεγονός ότι η Ιταλία δεν έχει υπογράψει την δικαστική συνεργασία, αλλά σίγουρα αυτή η παράληψη όσο και αν ζητάτε από αυτήν την ανακοίνωση, μπορούμε να... Εμεί να παροτρύνουμε την Ιταλία να το συνυπογράψει όσο γίνεται συντομότερα, αλλά δεν είναι δυνατόν να φανταστεί κανείς ότι αυτή η σύμβαση θα λύσει το πρόβλημα. Εγώ πιστεύω ότι επί τη βάση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων που έχουν τα θεσμικά κοινοτικά όργανα σε σχέση με τα δικαιώματα των τόμων και των πολιτών σε ίση δίκη, σε τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα θεμελιώδη, ε, το χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της κοινότητας, ε, το γεγονός ότι έχουμε δικαίωμα για ένα σύστημα διαφανό και το δικαίωμα κάθε πολίτη να είναι ο πρωταγωνιστής για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικαστικού χώρου, η Κομίσιον δεν μπορεί λοιπόν να περιορίζεται σε τέτοιο είδους απαντήσεις, αλλά πρέπει να μας δώσει και περαιτέρω εξηγήσει και απαντήσεις. Δεδομένε τη ιδιαίτερη ευαισθησία του θέματος, νομίζω πως όχι απλά μπορούμε να ε, γράψουμε επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στον πρόεδρο Μπαρόζο αλλά και στον αντιπρόεδρο Σεύκοβιτς που ασχολείται ακριβώς με αυτά τα θέματα αλλά να δώσουμε σχετική επιστολή στην είπατε εκπρόσωπο Άστον για να ζητήσουμε την παρέμβασή της όσο αυτό εμπίπτει στην αρμοδιότητές της να παρέμβει λοιπόν προς τις χώρες που εμπλέκονται στην υπόθεση και που προφανώς δεν εκφράζουν αυτή, πλήρως αυτή την ε, κοινοτική αλληλεγγύη στην οποία όλοι έχουμε συνυπογράψει από τη στιγμή που συμμετέχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούμε λοιπόν να αφήσουμε ανοιχτή αυτή την αναφορά και να ξεκινήσουμε αυτή τη διαδικασία επικοινωνίας με την Επιτροπή, τον Επίτροπο και την ε, είπατε εκπρόσωπο Άστρο. Σας ευχαριστώ και πάλι για την συμμετοχή σας και περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης που είναι η παριθμόν 14, η παριθμόν 1347 του 2011 και έχει υποβληθεί από την ε, Σέλμα Γκυλιερμίνα Γκόμες Αγκούλο, Ισπανική Ιθαγένεια, σχετικά με το δικαίωμα πρόσβαση που αφορούν τη σύλληψη και εκτέλεση του πατέρα της κατά τον εμφύλιο πόλεμο της Ισπανίας. Η κυρία αυτή είναι παρούσα και σας δίνω το λόγο για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Ζητάω δικαιοσύνη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί στην Ισπανία δεν μου την προσφέρουν. Για κάποιον άνθρωπο ο οποίος ήταν καλός και δεν έκανε κακό σε κανέναν. Ευχαριστώ. θα μιλήσω κι εγώ, είμαι η κόρη της. Να σας εξηγήσω λιγάκι ποια είναι η ιστορία του πατέρα μου. Πολιτικός από το Σοσιαλιστικό Κόμμα σκοτώθηκε στην αρχή του εμφυλίου πολέμου στην Ισπανία. Ποτέ δεν μάθαμε ούτε πώς τον σκότωσαν ούτε που τον έθαψαν. Και αυτό ακριβώ είναι και το μεγάλο δράμα της μητέρας μου, ότι ποτέ δεν το έμαθε. Και μάλιστα ποτέ δεν τον γνώρισε γιατί γεννήθηκε αφού εκείνος πέθανε. Για πολύ καιρό λοιπόν προσπαθήσαμε να βρούμε αρχεία. Γράψαμε σε τόσα κέντρα αρχείων στην Ισπανία δεν μπορείτε να φανταστείτε. Βρήκαμε κάποια χαρτιά τα οποία σας ε, στείλαμε εδώ στην Επιτροπή αυτή. Κοιτάξτε, προσέξτε λίγο τις ημερομηνίε των εγγράφων αυτών. Τα έγγραφα αυτά αντικαθιστούν στη... σε ένα κομμάτι της ζωής του παππού μου αναφέρονται διάφορα πράγματα. Ότι πέθανε το 1936. Αλλά οι ημερομηνίες αυτές μιλάνε για το 1937, για το 1941, για το 1943. Ε, ε, τι καταλαβαίνετε εσείς από αυτό. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος από ό,τι φαίνεται σκοτώθηκε και θάφτηκε σε ένα κοινό τάφο και για τον οποίο δεν έχουμε καμιά πληροφορία. Οι στρατιωτικές αρχές όμως και οι δικαστικές αρχές έχουν έγγραφα από το Δήμο στον οποίο απευθύνθηκαν για να ενημερωθούν για τα οικονομικά του στοιχεία αφού είχε πεθάνει. Κάτι το οποίο έχει συμβεί με όλα τα θύματα του, της εποχής του Φράνκο. Μετά το θάνατο δηλαδή ζητήθηκαν ε, τα ρέστα κατά κάποιο τρόπο από τον ε, παππού μου από το καθεστώς αυτό. Το ξέρανε δηλαδή ότι είχε πεθάνει και κάπου είχαν στοιχεία γι' αυτόν. Το τελευταίο έγγραφο είναι του 1943. Ένα έγγραφο από την επίσημη εφημερίδα της Κόρδοβα. Εκεί ο Δήμος της Ποσάδας λέει ότι τέσσερα χρόνια μετά τη λήξη του εμφυλίου πολέμου αρχιοθετήθηκε η υπόθεση. Τι έγινε όμως. Δεν μάθαμε ποτέ. Αυτή είναι η εμπειρία που έχουμε μέχρι τώρα. Γι' αυτό και εμείς ζητάμε περισσότερες πληροφορίες από το δικαστήριο της ε, Ποσάδας που δεν έκανε τον κόπο ποτέ να μας απαντήσει. Άλλα αρχεία απάντησαν, είτε ότι έχουν είτε ότι δεν έχουν αρχεία. Αλλά ο Δήμος της Ποσάδας, που εκεί έλαβαν χώρα τα γεγονότα, δεν μας απάντησε ποτέ. Για μας αυτό δείχνει έλλειψη σεβασμού και γι' αυτό είμαστε εδώ, γιατί πιστεύουμε ότι έχουμε δικαίωμα στην ενημέρωση, δικαίωμα στην πρόσβαση στην πληροφόρηση. Ε, συγγνώμη που σας ε, μιλάω έτσι, αλλά βλέπετε η απάντηση που έχουμε πάρει και έτσι καλώς σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούτε και που μας προσκαλέσατε να έρθουμε εδώ και να σας παρουσιάσουμε τη θέση μας η Κομισιόν τι μας λέει μας λέει ότι το δικαίωμα στην πληροφόρηση είναι κάτι προσωπικό δηλαδή δεν μπορεί ένας τρίτος να το ζητήσει συγγνώμη αλλά το δικαίωμα στην πληροφόρηση είναι το δικαίωμα στην πληροφόρηση για έναν πατέρα νεκρό εδώ και 66 χρόνια τι άλλο δικαίωμα δηλαδή μπορεί να υπάρχει πιο σημαντικό από αυτό δεν πλήττουμε τα προσωπικά δεδομένα κανενός, αντίθετα. Όταν δεν ξέρει κανεί πού είναι θαμμένα τα κόκαλα του πατέρα του, δεν θα έπρεπε να έχει δικαίωμα να το μάθει. Γι' αυτό και βρισκόμαστε εδώ. Και τρία-τέσσερα συγκεκριμένα πράγματα έχουμε να σα ε, πούμε. Ότι η Ισπανία δεν έχει μάλλον ακόμα συνυπογράψει την εισδοχή της στην ε, συμφωνία για πρόσβαση στα αρχεία. Είναι όμως κάτι πολύ βασικό για τις οικογένειες όλων των θυμάτων που βρίσκονται στην ίδια περίπτωση με την δικιά μου την οικογένεια και που αγνοούν πλήρως τι έχει συμβεί με τους δικούς τους. Όλοι θα έπρεπε να ακολουθούν την ίδια πολιτική απέναντι στις οικογένειες των θυμάτων, να τους ημερώνουν δηλαδή. Έπειτα θέλουμε να ζητήσουμε από το Δήμο της Ποσάδας να συνεργαστεί με την οικογένειά μας. Είναι έγγραφα τα οποία πρέπει να υπάρχουν ακόμα. Να τα ψάξουν παρακαλώ. Εμείς θέλουμε να ξέρουμε πού έχει θαυτεί ο παππούς μου. Τρίτον, η Ισπανία θα έπρεπε να έχει ε, μια τράπεζα ε, ADN DNA δηλαδή, όπου να μπορούν να παίρνονται δείγματα και να μπορούν έτσι να βοηθηθούν οι οικογένειες των θυμάτων και η μητέρα μου για παράδειγμα να μπορέσει να νιώσει καλύτερα. Γι' αυτό και σας ζητάω να μην κλείσετε αυτήν την υπόθεση παρακαλώ. Δεν θα ήθελα να πεθάνει η μητέρα μου χωρίς να ξέρει που έχει ταφεί ο πατέρας της. Είναι πιστεύω μια βοήθεια την οποία εσείς μπορείτε να προσφέρετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ ο Βίνσεντ Ντεπίν από την Κομισιόν. Thank you very Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι εννοείται ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα. Δημιουργεί αίσθηση. Το αντιλαμβανόμαστε αυτό πάρα πολύ καλά. Όμως, βλέπετε, εμείς αυτό που μπορούμε να απαντήσουμε είναι τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχουν λοιπόν ε, δεδομένα βάσει της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας που να επιτρέπουν σε μας να δώσουμε συνέχεια στο αίτημα ε, της αναφέρουσας. Η αναφέρουσα βασίζεται ε, σε διάφορα νομικά κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για παράδειγμα οδηγία 9546 για τα προσωπικά δεδομένα ή στην απόφαση του Συμβουλίου του 2008 για παράδειγμα 977 και αυτά τα δύο νομικά κείμενα ε, σαφώς ρυθμίζουν τη διαδικασία και την πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα. Αλλά όπως λέμε και εμείς στην απάντησή μας, αυτό έχει να κάνει με δεδομένα τα οποία είναι καθαρά προσωπικά, δηλαδή που αφορούν ε, το άτομο του οποίου τα προσωπικά δεδομένα επεξεργάζονται. Δεν μπορεί δηλαδή κάποιο να ζητήσει για κάποιον τρίτο. Ό,τι δεσμούς και αν έχει με αυτά τα άτομα, τα προσωπικά δεδομένα, έτσι όπως καθορίζονται από τα νομικά κείμενα, έχουν να κάνουν με τον άμεσα ενδιαφερόμενο. Ο ίδιος δηλαδή ο άνθρωπος μπορεί να ζητήσει πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα, αλλά όχι σε κάποιο άλλο. Λυπούμαστε που έχουν έτσι τα πράγματα, αλλά έτσι έχουν τα πράγματα. Οπότε βάσει αυτής της νομικής κατάστασης εμείς δεν μπορούμε να δώσουμε άλλη ερμηνεία χωρίς να παραβιάσουμε τους νόμους. Ένα άλλο στοιχείο που λέει η αναφέρουσα είναι ε, τα θεμελιώδη δικαιώματα, προστασία στην ε, αξιοπρέπεια, Αναφέρεται δηλαδή στα θεμελιώδη, στο χάρτη θεμελιωδιών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φυσικά τα δικαιώματα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά και διασφαλίζουμε την προστασία τους βάσει της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Υπενθυμίζω όμως ότι οι διατάξεις του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων έχουν να κάνουν μόνο με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και εφαρμόζονται μόνο όταν έχουμε να κάνουμε με μια Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Ενώ στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως είπα και στην αρχή, δεν υπάρχει καμία βάση στο ευρωπαϊκό δίκαιο που να μας επιτρέπει να προχωρήσουμε με αυτήν την δύσκολη υπόθεση. Σημειώσαμε όμως από το Συμβούλιο της Ευρώπης δεν είναι βέβαια αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έτσι είμαστε δύο εντελώ ε, διαφορετικά πράγματα, το Συμβούλιο της Ευρώπης ή το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και εμείς. Σημειώσαμε όμως ότι έχει υπάρξει ε, νομολογία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δεν είναι Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα δώσει συνέχεια ή θα αποφασίσει κατά πόσο το θέμα που εξετάζουμε εδώ είναι θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή όχι, αλλά να ξέρετε ότι έχει υπάρξει υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ε, για μια αντίστοιχη περίπτωση και ίσως εκεί να πρέπει να ε, αποφανθεί, να αποτανθεί συγγνώμη, η αναφέρουσα χωρίς φυσικά να προκαταλαμβάνουμε με τίποτα την απόφαση που θα πάρει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που όπως είπαμε είναι ξεχωριστό σώμα από εμά. Ευχαριστούμε κύριος Γιάννητς. Ευχαριστώ Πρώτα απ' όλα, σας ευχαριστώ και σας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις υπηρεσίες της Επιτροπής μας που έκαναν αποδεκτή την αναφορά αυτή. Αν κοιτάξουμε λίγο την ιστορία της χώρας μου τα 70 τελευταία χρόνια και κοιτάξουμε και την ιστορία της Επιτροπής αυτής, είναι θαύμα τελικά που έφτασε εδώ μία από τις ε, χιλιάδες περιπτώσεις αγνοωμένων από την περίοδο του φραγκισμού. Πολλά τέτοια δράματα υπάρχουν. Το ότι έφτασε εδώ μια απο τις χιλιαδες περιπτωσεις αγνοουμενων απο υπόθεση είναι φοβερό. Και όχι από κάποιον ευρωβουλευτή μάλιστα, ένας απλός άνθρωπος έρχεται εδώ και λέει πού είναι τα οστά του πατέρα μου ή του παππού μου. Είναι πραγματικό θαύμα. Γι' αυτό και ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις υπηρεσίε τη που αυτό το θέμα έχει φτάσει στην Επιτροπή μας. Μακάρι να μπορούμε να προχωρήσουμε και να βοηθήσουμε. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερον, ευχαριστώ και αναγνωρίζω την προσπάθεια που γίνεται από την Σέλμα και την Νοέλη, γιατί καταλαβαίνω ότι για αυτές είναι μεγάλη προσπάθεια να έρθουν και να φέρουν εδώ το θέμα τους, που είναι ένα θέμα τόσο προσωπικό και τόσο συναισθηματικό. Μακάρι βέβαια να μπορούσαν να μάθουν και ποιος δολοφόνησε τον δικό τους άνθρωπο, πότε, πώς και μιλάω για δολοφονία γιατί δεν πρόκειται για εκτέλεση. Γιατί εκτέλεση έχουμε όταν έχει προηγηθεί δικαστική απόφαση. Αλλά εδώ δεν υπάρχει κανένα έγγραφο που να δείχνει ότι υπήρξε κάποια δικαστική απόφαση. Άρα πρόκειται για δολοφονία. Λοιπόν, μέσω του DNA, μέσω άλλων στοιχείων, άμεσα ή έμεσα, καλό θα ήταν να, μπορούσα, να μπορούσε η οικογένεια να έχει πρόσβαση στα αρχεία αυτά στα οποία αναφέρθηκε για να βγάλει κάποιο συμπέρασμα και να μπορέσει να τον θάψει με αξιοπρέπεια. Θα ήθελε βέβαια πολύ η οικογένεια να ε, καταδικαστούν και να τιμωρηθούν και υπεύθυνοι της δολοφονίας αυτής, που μάλλον έχουν βέβαια πεθάνει και αυτοί. Στα αρχεία λοιπόν που έχουν κλείσει, καλό θα ήταν να ανοίξουν για να βρεθούν στοιχεία τα οποία θα οδηγήσουν κατά πάσα πιθανότητα σε στοιχεία όπως αυτά που θέλει η οικογένεια. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το στηρίξουμε. Και μια ακόμα παρατήρηση θέλω να κάνω. Δεν είναι μόνο θέμα εσωτερικής πολιτικής της Ισπανίας. Εννοείται η σημερινή Ισπανία δεν φταίει, δεν έχει να κάνει ούτε με τους σοσιαλιστές, ούτε με το Ισπανικό Λαϊκό Κόμμα. Όλα αυτά είναι άλλο πράγμα, έτσι. Μιλάμε εδώ πέρα τώρα για ιστορική δικαιοσύνη, την οποία ε, κουβαλάνε στους ώμους τους οι οικογένειες, τα παιδιά, που έχουν υποφέρει από τις ε, εξαφανίσεις αυτές των δικών τους. Γι' αυτό και λέω ότι πρέπει να τους στηρίξουμε και να τους βοηθήσουμε, να προσπαθήσουμε να ικανοποιήσουμε το αίτημά τους όσο μπορούμε περισσότερο. Υπάρχουν χιλιάδες μελέτες ψυχολογικές, ψυχιατρικές και κοινωνικές για το πένθος. Αν δεν υπάρχει πτώμα, δεν μπορεί να πενθήσει ο συγγενής. 70 χρόνια μετά τον έχει το θάνατο μέσα τη οικογένεια σαν να προέκυψε χτες. Δεν έχει μπορέσει να πενθήσει, να περάσει από τη διαδικασία του πέντρου. Αυτό είναι τρομερό. Είναι κάτι το οποίο εμείς οι Ισπανοί, οι πολιτικοί το καταλαβαίνουμε, το αναγνωρίζουμε. Και είναι αλήθεια ότι δεν κάναμε ό,τι θα έπρεπε να είχαμε κάνει παρά τις προσπάθειες που μπορεί να έκανα διάφορες προσπάθειες ή το κοινοβούλιο. Τελικά δεν έχουμε κάνει αρκετά. Γιατί σύμφωνα με μια σοβαρή έρευνα του δικαστή Καρθών 114 άτομα που ήταν αγνοούμενοι εντοπίστηκαν τελικά από τους χιλιάδες και χιλιάδες. Είναι ο μεγαλύτερος αριθμός μετά την Καρπότζα, Πολ Πότ θυμηθείτε. Οι αρχές συμπεριλαμβάνουν και τον εαυτό μου σε αυτές, έτσι. Δεν μπορέσαμε να ικανοποιήσουμε το αίτημα των οικογενειών των αγνοούμενων αυτών που θέλουν να μάθουν τι έχει γίνει με τους δικούς τους. Η πρώτη απάντηση είναι αρνητική από ό,τι έχω δει. Εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι το συμπέρασμα της Κομισιόν. Το συμπέρασμα που είναι πάρα πολύ σύντομο και τι λέει. Λέει Μιλάει για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ότι θα μπορούσε να πάει εκεί η οικογένεια. Γιατί στην περίπτωση Γιάννο Βιέτς, που είναι η περίπτωση του Κατίν, έτσι, της ε, του Κατίν, λέει ότι όταν ένα κράτος δεν είναι νομικά υπεύθυνο για το θάνατο ή την εξαφάνιση ενός ατόμου, βάσει του άρθρου 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, πρέπει να επιδεικνύει στάση συμπόνιας και σεβασμού Συμπόνια και σεβασμό λοιπόν όσον αφορά την αγωνία των συγγενών θανόντων ή εξαφανιστέντων προσώπων και να βοηθά τους συγγενείς να συλλέγουν πληροφορίες και να αποκαλύπτουν τα συναφή γεγονότα. Και μετά λέει η σιωπή των κρατικών αρχών ενώπιον των πραγματικών <coughs> ανησυχιών των συγγενών μπορεί να χαρακτηριστεί μόνο ως απάνθρωπη συμπεριφορά τα λέει όλα. Όλοι είμαστε υπέρ των διεθνών συμβάσεων ε, του ΟΗΕ ε, και λοιπά για τις, την κακή μεταχείριση. Λοιπόν, κάποιο δικαστήριο είπε ότι τελικά συμπεριφερόμαστε απέναντι στα θύματα απάνθρωπα. Γι' αυτό επιμένω ότι πρέπει να δείξουμε ανθρώπινη συμπεριφορά και έτσι η Επιτροπή μας να γράψει ιστορία με την υπόθεση αυτή και να δικαιώσει, να στηρίξει το αίτημα της αναφέρουσας για να μάθουν οι κόροι και οι εγγονοί του αποθανόντος να μάθει περισσότερα πράγματα. Ήταν από το σεσολιστικό κόμμα, να, η φωτογραφία του για να μπορέσει να αναπαυθεί εν ειρήνη επιτέλους. Ευχαριστούμε κύριος Μέγερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να αναφερθώ στις δύο αναφέρουσες και να τους πω ότι εγώ προσωπικά ε, φόρο τιμής στον πατέρα και παππού τους. Ξέρω ότι υπάρχουν χιλιάδες και χιλιάδες οικογένειες στην Ισπανία που είναι αντιμέτωπες με το ίδιο πρόβλημα και που περιμένουν μία καλή απάντηση, μία διόρθωση κατά κάποιο τρόπο. Δεν είναι δυνατόν μετά τα γεγονότα και το τέλος του εμφυλίου πολέμου να είμαστε εδώ που βρισκόμαστε. Στην Ισπανία και σε... γλιτώσαμε από το φασισμό, σε άλλες χώρες έμεινε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δηλαδή, στην Ισπανία έμεινε, ενώ σε άλλε χώρε δεν υπήρχε πια. Συνεπώ, για τον Ανσέλμα Κυρμίνα Γόμε ε, Αγγούλο, για σας θέλω να σας πω ότι υπάρχει νόμιμη κυβέρνηση βέβαια στην ε, Ισπανία, η οποία θα έπρεπε να μπορεί να βοηθήσει. Και επίση να πω ότι είναι η πρώτη φορά που έρχονται τα γεγονότα αυτά εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όπω ε, είπε και ο συνάδελφος, χιλιάδες άλλοι σαν και εσάς αγνούν πλήρως που βρίσκονται τα οστά των δικών τους ανθρώπων που χαθήκαν είτε κατά τη διάρκεια του πολέμου είτε εκτελέστηκαν πολλές φορές εντελώς εξοδικαστικά απλώς και μόνο γιατί είχαν δημοκρατικές ιδέες. Γι' αυτό θέλω να πω ότι έχω κάθε σεβασμό απέναντί σας. Η αναφορά σας είναι πολύ σημαντική. Όχι μόνο για τον ε, πατέρα σας, ε, Δόνιαν Σέλμα, αλλά και για τον παππού σας, Δόνιαν Έλα, αλλά και γιατί είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να λυθεί στην Ισπανία. Με τον νόμο για την ιστορική μνήμη, σε ένα βαθμό λύθηκε, δεν είναι βέβαια αρκετό, δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει λυθεί το μεγάλο αυτό πρόβλημα, ούτε ότι έχει υπάρξει αποκατάσταση για όλους αυτούς τους ανθρώπους που αδικήθηκαν. Το δικό σας το αίτημα πάντως σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δείχνει ότι όλες οι δημόσιες δικήσεις πρέπει να βοηθήσουν για να υπάρξει ενημέρωση και αποκατάσταση. Οπότε από τη δικιά μου την πλευρά να ξέρετε ότι σας στηρίζω προκειμένου να τα καταφέρετε. Δεν θα σταματήσουμε να προσπαθούμε για να έχετε όλες τις πληροφορίες που θέλετε. Είναι πληροφορίες που πρέπει να τις έχετε. Τώρα, όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κοιτάξτε, είναι ένα θέμα που πηγαίνει πέρα από τις ε, όποιες ρυθμίσεις, εννοείται. Θέλεγα, λοιπόν η πρόεδρος της Επιτροπής μας να στείλει μια επιστολή στα δύο δικαστήρια τα οποία δεν σας βοήθησαν με πληροφορίες. Η πρόεδρός μας, στην Ισπανία δηλαδή, να απευθυνθεί σε αυτούς τους δύο δήμους, στις δικαστικές αρχές, εκεί προκειμένου να σας δώσουν τις πληροφορίες που θέλετε. Να περιμένουμε την απάντησή τους και στο μεταξύ να μείνει η αναφορά αυτή ανοιχτή, να μην κλείσει. Έτσι ώστε να παρακολουθήσουμε την υπόθεση και να προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο αδιαφυσβήτητες, έτσι, τακτικές. Να φροντίσουμε να πάρετε τις πληροφορίες που θέλετε, γιατί είναι δίκαιο. Τις δικαιούστε. Η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανοίγει κάποια πόρτα για παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να έρθουν από άλλα όργανα. Από τη δικιά μας την πλευρά πάντως, επειδή το αίτημά σας είναι ιστορική σημασίας, Πιστεύω ότι η αναφορά αυτή πρέπει να παραμείνει ανοιχτή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρακολουθήσουν την υπόθεση έτσι ώστε να πάρετε όλες τις πληροφορίες που θέλετε. Είναι σημαντικές φυσικά για σας και για τις οικογένειές σας, αλλά είναι σημαντικές και για το σύνολο της ισπανικής κοινωνίας, αλλά και της ευρωπαϊκής μάλιστα θα έλεγα, γιατί μιλάμε για τις συνέπειες ενός φασιστικού πραξικοπήματος. Οι άνθρωποι οι οποίοι αντιστάθηκαν σε αυτό το καθεστώς είναι άνθρωποι που αξίζουν το σεβασμό μας και αξίζουν την προσπάθεια αυτή που προτείνω για να παραμείνει ανοιχτή αναφορά. Ευχαριστώ, ε, κύριος Ρωμεβά. Σας ευχαριστώ. Συμφωνώ στις ευχαριστίες προς την Επιτροπή που έχει δεχτεί την αναφορά αυτή. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τις αναφέρουσες για τα λόγια τους, την κόρη δηλαδή και την εγγονή. Είναι πολύ βασικό το θέμα αυτό, αν μη τι άλλο, να παραμείνει ανοιχτό. Μέχρι να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε θετικά σε αυτό που μας ζητάνε. Δύο πράγματα εμένα μου κάνουν εντύπωση. Το ένα είναι αυτό που διάβασα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την επιχειρηματολογία της ε, δηλαδή όσον αφορά την προσφυγή ε, στην ε, προστασία προσωπικών δεδομένων που λέει ότι εδώ δεν στέκει. Για μένα είναι πολύ δύσκολο να το πούμε αυτό. Πόσο μάλιστα για τις οι οικογένειες που τι μαθαίνουν, μαθούν ότι δεν έχουν δικαίωμα να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα ενός ατόμου το οποίο ε, δεν μπορεί από μόνο του να τα ζητήσει αφού δεν υπάρχει. Οπότε, εμένα αυτό δεν μου φαίνεται πολύ σοβαρό σαν επιχείρημα. Αυτό είναι το ένα. Γι' αυτό και συμφωνώ με την ε, πρόταση των συναδέρφων να παραμείνει ανοιχτή αναφορά. Στηρίζω επίση και αυτό που είπε ο κύριο Μέγερ, δηλαδή να σταλούν αυτέ οι δύο επιστολέ από την Πρόεδρό μα στι αρμόδιε αρχέ τη Ισπανία για να ζητήσουμε να δοθούν οι πληροφορίε που ζητούν οι αναφέρουσε. Έχω όμω και ένα τρίτο στοιχείο να προσθέσω εδώ. Είναι σημαντικό Τη στιγμή που το μόνο που ζητάνε οι αναφέρουσε είναι πληροφορίε, να υπενθυμίσουμε ότι μετά από τόσα χρόνια δημοκρατία στην Ισπανία, το θέμα είναι δυνατόν έπρεπε να φτάσει μέχρι εδώ. Τι σημαίνει αυτό. Αυτό σημαίνει ότι οι μηχανισμοί οι οποίοι υπάρχουν ώστε να φτάσουμε στην αποκατάσταση δεν φτάνουν, δεν είναι αρκετοί ή δεν λειτουργούν καλά. Θα έπρεπε λοιπόν να στείλουμε και αυτό το μήνυμα κατά τη γνώμη μου, να πετήσουμε δηλαδή από τις αρμόδιες αρχές τέτοιου είδους περιπτώσεις, αν μη τι άλλο, αν μη τι άλλο, να τις ακούνε, να τους δίνουν προσοχή. Τέλος, κάτι συγκυριακό άλλο νομίζω ότι είναι σημαντικό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει από την αναφέρουσα να πάει σε εθνικές αρχές. Μα μόνος δικαστής μέχρι τώρα που έχει παρακολουθήσει τέτοιες ε, περιπτώσεις ήταν θύμα μιας ε, εκστρατείας δυσφήμισης σε βάρος του. Καταλαβαίνετε ότι και αυτό μου φαίνεται ιδιαίτερα ανησυχητικό. Γιατί, γιατί ακριβώς αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο δικαστής προσπάθησε να κάνει αυτό ακριβώς που ζητούν οι αναφέρουσες στην Ισπανία. Αφού λοιπόν έφτασε εδώ η συζήτηση, σας λέω πρώτον είναι ανησυχητικό γιατί αυτό σημαίνει ότι δεν μπόρεσε να λυθεί προηγουμένως τους μηχανισμούς που έχουμε πριν από εδώ και γι' αυτό δεν θα έπρεπε να κλείσει η αναφορά αυτή. Ευχαριστούμε κυρία Όκεν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να συμφωνήσω με αυτά τα οποία ακούστηκαν. Πρώτα απ' όλα βεβαίως ευχαριστώ την οικογένεια που ήρθε εδώ πέρα και τους συναδέλφους αλλά πραγματικά απορώ με τα επιχειρήματα της Κομισιόν. Είναι ντροπή νομίζω να, να, να προσφέρει τέτοια αντίστροφα επιχειρήματα. Δηλαδή υπάρχει ένα, ένας νόμος ο οποίος χρησιμοποιείται τελικά για ποιο λόγο. Για να προστατευτούν οι αρχές από τους ανθρώπους και όχι αντιστρόφως. Οπότε να πω πως Σπάνια έχω διαβάσει κάτι τόσο ανησυχητικό όσο αυτή εδώ πέρα η δικαιολογία ότι είναι προσωπικά δεδομένα. Μα τι προσωπικά δεδομένα, ο άνθρωπος εξαφανίστηκε. Και μάλλον τον, τον εκτέλεσαν. Έχουμε το δικαίωμα εμείς να ασχοληθούμε με κάτι το οποίο έρχεται ενώπιον μας. Είμαστε πολιτικοί. Δεν είναι ανάγκη να κοιτάμε το τι μπορεί να σταθεί ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Εάν ε, ε, είναι επιτρεπτή μια αναφορά, πρέπει να την εξετάσουμε. Και αν μ' ακούει κανείς, δύο λόγια προς την Ισπανική κυβέρνηση. Εάν θέλει κανείς συμφιλίωση, που προφανώς ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί στην Ισπανία, μετά από τόσα χρόνια, ε, πρέπει να, να μαθευτεί η αλήθεια. Το ξέρουμε και από άλλα μέρη του κόσμου, όπου υπήρξε συμφιλίωση μετά από μεγάλες συγκρούσεις. Τρία σημεία λοιπόν περιέχει η ε, συμφιλίωση. Δικαιοσύνη, ειρήνη και την ε, αλήθεια. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν μετά από τόσα χρόνια δημοκρατίας στην Ισπανία να υπάρχουν δυνάμεις που προσπαθούν να αποκρύψουν την αλήθεια. Και αυτό σημαίνει πως υπάρχουν ακόμα ε, μεγάλα χάσματα, σχίσματα στην ισπανική κοινωνία. Και εμείς ως εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να φροντίσουμε και οι Ισπανοί πολίτες να, να νιώσουν ότι το να είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει πως τώρα ε, πραγματικά ε, γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν είναι. Δεν υποτίθεται πως ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα υπερισχύουν όλων των άλλων. Θέλω η Κομισιόν να κάνει σωστά τη δουλειά της εδώ πέρα και δεν την έχει κάνει σωστά εδώ πέρα. Πρέπει λοιπόν να κρατήσουμε ανοιχτή αυτή την αναφορά και να απευθυνθούμε στην Ισπανία και να ζητήσουμε να ξεκαθαρίσει αυτή η υπόθεση. Και είναι ξεκάθαρες νομίζω και οι αποφάσεις του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. να γράψουμε μια επιστολή, να βάλουμε το όνομά μας από κάτω, να τη στείλουμε στην Ισπανία και να πούμε κοιτάξτε τι έχει ήδη αποφασίσει για ανάλογες περιπτώσεις το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Και οι Ισπανοί ούτως ή άλλως θα βρουν τη λύση. Είπε και το δικαστήριο του Στρασβούργου πως είναι απάνθρωποι αυτή η συμπεριφορά και δεν είναι δυνατό να υπερασπιζόμαστε τέτοια απάνθρωπη συμπεριφορά με νομικίστικες ε, εξυπνάδες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής είπε ότι είναι ένα ευαίσθητο θέμα που δημιουργεί η αίσθηση. Όλα αυτά τα θέματα όντως είναι πολύ ευαίσθητα. Τώρα πριν μπω στην ουσία της αναφοράς, θα ήθελα να σας πω πού ακριβώς βρισκόμαστε εδώ στην Επιτροπή αυτή αναφορών. Γιατί εμείς που είμαστε εδώ πολύ καιρό, όπως ο Μιχαήλ Άγχελ Μαρτίνες για παράδειγμα, ξέρουμε τι γίνεται όταν έχουμε τέτοια θέματα. Η κυρία Οκέ λέει στους Ισπανούς συχνά «Σκεφτείτε περισσότερο ευρωπαϊκά και λιγότερο ισπανικά». Πώς όμως να μην σκεφτεί κανείς ισπανικά Μάργαρετ, μην εκνευρίζεσαι, μην εκνευρίζεσαι. Μα το λέω αστιαβόμενος. Γιατί υπάρχουν ένα σωρό άλλα θέματα. Μάργαρετ, μην το παίρνει έτσι. Εσύ μας λες ότι οι Ισπανοί όλο μιλάμε, όλο φωνάζουμε και ότι πρέπει να σκεφτόμαστε πιο πολύ ευρωπαϊκά. Ε, ναι, δεν ξέρω αν δεν στο μετέφρασαν καλά ή δεν κατάλαβες. Εγώ δεν επιτέθηκα εναντίον σου. Αντίθετα, Μάργαρετ, αυτό που είπα ήταν θετικό για σένα. Ότι μερικές φορές πρέπει να σκεφτόμαστε όντω πιο ευρωπαϊκά. Αυτό λέω. Μην πετάς λοιπόν το στυλό στο ταβάνι και άκουσέ με για να με καταλάβεις. Λέω λοιπόν ότι είναι μια ιστορική στιγμή για την Επιτροπή Αναφορών σήμερα δεν είναι όπως έλεγε και ο Λουίς, δεν είναι θέμα δεξιάς, αριστεράς, σοσιαλιστών και δεν ξέρω εγώ τι. Όχι. Στον 20ο αιώνα στην Ευρώπη έχουμε περάσει από τόσες αντιπαραθέσεις, τόσους πολέμους. Σήμερα ας ανοίξουμε μια πόρτα. Όταν έρχονται συγγενείς και από τον πρώτο και από τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ε, για τους αγνοούμενους στην Κύπρο, ή άλλοι από την ε, Κροατία με τον πόλεμο στα Βαλκάνια ή από την Ανατολική Ευρώπη, την πόρτα να τους την ανοίγουμε. Και το κάναμε. Την ανοίξαμε μέχρι τώρα αυτή την πόρτα εμείς στην Επιτροπή Αναφορών σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που ήθελαν να έχουν νέα για τους δικούς τους. Από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ε, έχω κάτι που απάντησαν στην αναφέρουσα. Η προηγούμενη κυβέρνηση του Ροντρίγκε Σταποτήρο το 2011, πριν από τη σημερινή δηλαδή κυβέρνηση του Μαριάνο Ραχόη, ζητήθηκε ή προσπαθήσανε μάλλον να βρούνε ίχνη για όλους αυτούς τους αγνοούμενους, που είναι στην ίδια περίπτωση όπως και ο πατέρας σας. Εστάλει επιστολή λοιπόν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για τα προβλήματα τα οποία οι προσπάθειες για να βρεθούν ε, στα αρχεία τα διάφορα έγγραφα, αν δεν απατώμε, περάσανε από την Κόρτοβα στην ε, Ποσάδας, από το Ποσάδα στην Κόρτοβα, στο Περιφερειακό Αρχείο εκεί. Όλες οι προσπάθειες που έγιναν έμειναν χωρίς αποτελέσματα σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τις κυβερνήσεις οι οποίες ε, είχαν την ευθύνη της περιφερειακές κυβερνήσεις, τέλος πάντα που είχαν την ε, ευθύνη. Το ίδιο το Υπουργείο Δικαιοσύνης λέει ότι για τέτοιες περιπτώσεις όπου δεν μπόρεσαν να βρεθούν τα έγγραφα που ζητούνται, δεν ξέρουν αν κάηκαν, αν εκλάπησαν, αν καταστράφηκαν δεν μπορούν να τα βρούνε παρά το γεγονός ότι ζητήθηκαν, ε, προσοχή, παρά το γεγονός ότι ζητήθηκαν, λέει. Αυτό το λέει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, έτσι. Για το δεύτερο το οποίο λέτε στην αναφορά σας. Γνωρίζετε ότι η αρμοδιότητα για να ζητήσει κανείς την εκταφή και την αναγνώριση Την αρμοδιότητα την έχει ο Δήμος της Κόρδοβα και η αυτόνομη περιφέρεια της Ανδαλουσίας. Συνεπώς, πρέπει να καταλάβουμε ότι το θέμα των αρχείων και αρμοδιότητα της εκταφής είναι αρμοδιότητες μιας αυτόνομης περιφέρειας, που είναι η Ανδαλουσία σε αυτή την περίπτωση. Οπότε σε αυτούς πρέπει να πούμε και να υπενθυμίσουμε. Όπως είπαν και προλαλήσαντες εδώ που είναι τα κόμματά τους, πας που έχουν και τα ενία στην Ανδαλουσία. Δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι οι δύο συνάδελφοι που είναι από εκεί θα προωθήσουν το θέμα ώστε το Υπουργείο Δικαιοσύνης να δώσει κάποια συνέχεια. Δεν θέλω να δώσουμε την εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν κάνει ας πούμε, καλά τη δουλειά της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι δεν είναι αρμόδιοι. Επιστολές όμως μπορούμε να στείλουμε. Οπότε, εσείς είπατε να στείλουμε επιστολές στην δικαιοσύνη. Μα η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη. Στη δικαιοσύνη δεν μπορούμε εμείς να πούμε τι πρέπει να κάνει. Δεν πρέπει να απευθυνθούμε στη δικαιοσύνη γιατί έχουμε να κάνουμε με μια περίπτωση που όλοι οι πολιτικοί οι δημοκρατικοί εδώ γνωρίζουμε ότι η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη. Ξέρει τι αποφάσεις να πάρει. Αυτές τις επιστολές πρέπει να τις στείλουμε στις αρχές, τις πολιτικές αρχές που συνδέονται με κάποιο τρόπο με το θέμα. Εφόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα γιατί δεν είναι αρμόδια για την υπόθεση αυτή, να ζητήσουμε από την Περιφερειακή Κυβέρνηση της Ανδαλουσίας και από το Δήμο της Κόρδοβα και από τα αρχεία, σε αυτούς να στείλουμε επιστολή. Έτσι λέω εγώ, κυρία Πρόεδρε. Και ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι εδώ βρισκόμαστε μπροστά σε μια σοβαρή υπόθεση η οποία όντως μας βάζει μπροστά στις ευθύνες μας και βάζει τους ε, ευρωβουλευτές μπροστά στις ευθύνες τους. Ο Γέρμο Κανούντες που σίγουρα από κάπου ψηλά θα μας ακούει, θα ευχαριστεί την οικογένειά του που έφερε το θέμα του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και εμείς πρέπει να ευχαριστήσουμε την οικογένειά του που έκανε το βήμα αυτό. Έκανε μια τεράστια προσπάθεια και θυσία για να φέρει την υπόθεση εδώ προς συζήτηση. Δεν είναι απλό πράγμα, είναι μια προσωπική υπόθεση που έχει βέβαια μεγάλη αξία και ως προσωπικό θέμα, αλλά επιπλέον είναι ευρύτερο, ξεπερνάει τα όρια του ατόμου. Αναπόφευκτα. Γιατί αφορά πολλούς ανθρώπους, άρα είναι και συλλογικό. Και αυτό το είπαν και οι συνάδελφοι εδώ όλοι όσοι πήραν το λόγο μέχρι τώρα. Και όλοι οι Γιάννης και ο Ρουντιμέγερ και ο Ρωμέβα. Α, και ο Τουρκάης. Ναι. Όλοι, όλοι το είπανε. Όλοι το αναγνωρίζουμε ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια στιγμή πολύ σημαντική που ανοίγει μία πόρτα. Και είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να κάνει ένας ευρωβουλευτής, να ανοίγει μία πόρτα στις διεκδικήσεις για την εφαρμογή και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ανοίγει μια πόρτα λοιπόν εδώ για να ακούσουμε και να καταλάβουμε τη φωνή χιλιάδων και χιλιάδων πολιτών των οποίων παραβιάστηκε ένα πολύ βασικό δικαίωμα ε, που έχουν στη ζωή τους για χρόνια τους, ε, δεν τους αποκαλύφθηκε η αλήθεια, η ιστορία. Ε, λοιπόν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σήμερα και η Επιτροπή μας έχει την ευκαιρία να ανοίξει την πόρτα για να δοθεί λύση. Το ότι είναι συλλογικό το θέμα αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να βασιζόμαστε σε κάποια απλοϊκά επιχειρήματα. Αδύναμα μάλλον πιο σωστά επιχειρήματα. Εγώ πιστεύω ότι η Επιτροπή μας θα έπρεπε να ζητήσει επιπλέον νομικές ε, γνωματεύσεις σχετικά με το όσα μας λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επιπλέον λοιπόν νομικές γνωματεύσεις που να μας ενισχύουν στην πεποίθησή μας ότι μπορούμε να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των πολιτών, τα ανθρώπινα δικαιώματα και που να μπορούν να μας βοηθήσουν στο μέλλον να λύνουμε τέτοιες περιπτώσεις. Αυτό είναι κάτι επιπλέον δηλαδή που ζητάω πέρα από αυτά που ήδη ζητήσαμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την άλλη. Το είπαν και οι συνάδελφοι. Να αφήσει ανοιχτή την πόρτα, ανοιχτή την ανηφορά, ώστε να αναλάβει την ευθύνη να μην κλείσει, να μην σταματήσει αυτή η ιστορική σημασίας ε, εξέλιξη να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τις θέσεις μας και τελικά κανένας από όσους ήταν εδώ παρόντες, κανένας από την οικογένεια του Αντσέλμου Κογέρμου Κόμες Δεμούδες, ούτε κανένας άλλος από τους χιλιάδες αυτούς Ισπανούς που είναι θύματα της ίδιας κατάστασης να μην μείνουν χωρίς να προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματά τους το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή μας. Συμφωνώ λοιπόν με τα όσα είπαν και οι προλαλήσαντες εδώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μαρτίνες Μαρτίνες. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η αλήθεια είναι ότι ε, έχουν υποθεί περίπου όλα. Θέλω κι εγώ να πω ότι συμφωνώ με τους προλαλήσαντες. Και χαίρομαι πάρα πολύ που μίλησε και η κυρία Όκεν γιατί όντως δεν θα έπρεπε να είναι ένα θέμα καθαρά ισπανικό αυτό. Είναι πολύ σημαντικό στη συζήτηση αυτή να συμμετέχουν και άλλοι Ευρωπαίοι και άλλοι δημοκράτες. Θα ήθελα επίσης η οικογένεια να γνωρίζει ότι και ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παίρνει θέση και βουτάει στα βαθιά νερά όπως έκανα κι άλλοι συνάδελφοι εδώ. Πρώτα απ' όλα λοιπόν θέλω να υπογραμμίσω την ε, επιμονή της οικογένειας. Όντως πρόκειται για ένα φόρο τιμής όπως ακούσαμε. Είναι φόρος τιμής προς την οικογένεια η οποία το και η εγγονή του η οποία υπέφερε σε όλη της τη ζωή. Χωρίς να παραιτηθούν όμως, συνέχισαν πιστεύοντας σε, στα δημοκρατικά όργανα παρόλο που θα μπορούσαν κάλλιστα μετά από όλες τις δυσκολίες αυτές που αντιμετώπισαν είχαν παραιτηθεί. Αυτό μας αναγκάζει να πάρουμε θέση που δεν θα τους απογοητεύσει. Διότι ουσιαστικά δείχνουν ότι έχουν εμπιστοσύνη στην Ευρώπη της δημοκρατίας, στην Ευρώπη των αξιών εκείνων που ακριβώς είχαν σαν αποτέλεσμα η Ισπανία να μην μπορέσει από την αρχή να συμμετέχει στο ευρωπαϊκό δημοκρατικό αυτό σύστημα, αλλά να έρθει 30 χρόνια αργότερα. Συνεπώς, αν τους απογοητεύσουμε θα ήταν πάρα πολύ σοβαρό. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί είχαν την επιμονή, την, ε, το πείσμα, παρά τις δυσκολίες, να συνεχίζουν. Και έφτασαν εδώ. Το είπε ποιος ο Ντρουγάης νομίζω. Έφτασαν εδώ με ελπίδα, όχι μόνο να τους ακούσουμε, να τους ακούσουμε και στη συνέχεια να τους ανοίξουμε το δρόμο ώστε το αίτημά τους να μην θαυτεί όπως έτσι άσχημα θαύτηκε και παραμένει ο Ανσέλμο. Η συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν είναι μια ευρωπαϊκή περίπτωση. Είναι μια περίπτωση όπου η εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα μου, όπως και σε πάρα πολλές άλλες χώρες, ε, δεν βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση γιατί απομακρυνόμαστε μερικές φορές σε, από αξίες όπως είναι η αλληλεγγύη και η δημοκρατία. Γι' αυτό σήμερα είναι πάρα πολύ σημαντικό να απαντήσουμε με συνέπεια απέναντι στις αξίες αυτές. Τώρα η συγκεκριμένη υπόθεση έχει να κάνει, το είπε και Λουίς ε, Γιάννηθ πριν, έχει να κάνει με ένα αίτημα απλό που δεν μπορεί κανείς να γνωρίσει. Εδώ δεν μας ζητάνε τίποτα φοβερό. Είναι ένα θέμα ζωντανό. Και ζωντανό όχι μόνο όσο ζει η κόρη του που είναι της δικιάς μου γενιάς, αλλά και όσο ζει η εγγονή του, τα παιδιά της και τα εγγόνια της. Πρέπει να κλείσει καλά αυτή η υπόθεση και όχι άσχημα. Μέχρι τώρα δεν μπορέσαμε να βρούμε τη λύση που θέλαμε. Για τη συγκεκριμένη λοιπόν περίπτωση πρέπει να ξέρουμε ότι είναι μια περίπτωση που απαιτεί κάτι βασικό. Γι' αυτό και πρέπει να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά πρέπει να πάει στη νομική υπηρεσία. Και αντιλαμβάνομαι αυτά που λέει βέβαια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν πιστεύω ότι από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η απάντηση είναι «Α, ας το παρακάμψουμε». Όχι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε αυτό που έχουμε πει και άλλες φορές εδώ, ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη διάταξη στην κοινοτική νομοθεσία που να επιτρέπει να μιλήσουμε για παραβίαση. Εντάξει, αυτό το καταλαβαίνω. Αυτό όμως που παραβιάζεται είναι οι θεμελιώδεις αξίες και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι θεματοφύλακας των συνθήκων και οι συνθήκες είναι εκείνες που κάνουν τις θεμελιώδεις αυτές αξίες ακρογωνιαίο λίθο του Ευρωπαϊκού Οικοδομήματος. Συνεπώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αποπείται ευθυνών, εντάξει, πρέπει να λάβει υπόψη της ότι εμείς θέλουμε να συνεχίσουμε να αφήνουμε ανοιχτή την αναφορά για να βρούμε λύσεις στη συγκεκριμένη περίπτωση που μας απασχολεί. Και να διατηρήσουμε βεβαίως και ζωντανή την ελπίδα της παραδειγματικής αυτής οικογένειας. Έχω να σας πω δύο ακόμα πράγματα. Το ένα είναι, γιατί είναι το μόνο που δεν είπαμε μέχρι τώρα, είναι ότι είμαστε, έχουμε να κάνουμε με θύματα τρομοκρατίας. Οι δύο κυρίες που βλέπετε εδώ στην αίθουσα είναι δύο θύματα με όνομα και επίθετο της τρομοκρατίας. Όπως έχουμε θύματα από την τρομοκρατία, από άλλες τρομοκρατικές δραστηριότητες που γνωρίζουμε στην Ισπανία. Αν δεν δείξουμε την αλληλεγγύη μας προς αυτές, είναι σαν να μην δείχνουμε αλληλεγγύη ούτε σε άλλα θύματα τρομοκρατίας στην Ισπανία από τα πρόσφατα χρόνια μάλιστα. Τέτοια είναι η φύση του θέματος. Και το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι για να κάνει κανείς αυτοκριτική, γιατί είμαστε πολιτικοί πολλά χρόνια και ο Βίλη και ο Λουίς, όλοι όσοι είμαστε λίγο πολύ εδώ από την Ισπανία, άρα μπορούμε να κάνουμε και αυτοκριτική. Βλέπετε, στην Ισπανία δεν έχουν κλείσει πολλά θέματα. Εγώ ζω σε ένα δήμο που δεν είναι ένα χωριό, είναι μια πόλη. Και όταν κυκλοφορώ στο δρόμο, πηγαίνω, ε, βγαίνω το σπίτι μου και φτάνω σε ένα δρόμο που ονομάζεται ηλεοφόρος του Χενεραλίσιμο, όπως ονομαζόταν ο Φράνκο. Είναι σαν να ονομάζαμε λεωφόρο του Ντούτσε, λεωφόρο του Φίρερ. Αυτή είναι η λεωφόρος στην γειτονιά που ζω στη Μαδρίτη. Και υπάρχουν και πάρα πολλοί δήμοι που εξακολουθούν να έχουν δρόμους με τέτοια ονόματα. Οπότε μπορώ να φανταστώ πώς αισθάνονται οι γυναίκες αυτές όταν βρίσκονται σε τέτοια περίπτωση. Εγώ όταν βλέπω πώς λέγεται ο δρόμος αυτός, πραγματικά αρρωσταίνω. Πόσο μάλλον άνθρωποι που έχουν υποφέρει έτσι όπως έχουν υποφέρει οι δύο αυτές κυρίες. Στην Ισπανία λοιπόν εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν έχουν κλείσει και που θα έπρεπε να κλείσουν. Στην Δημοκρατική Γερμανία του σήμερα κανείς δεν μπορεί να φανταστεί ένας δρόμος να ονομάζεται ηλοφόρος του Φίρερ ούτε του Στάλιν. Ε, αυτή είναι η πραγματικότητα όμως μέσα στην οποία ζούμε εμείς στην Ισπανία, σε, πολλές, ε, σε πολλούς δήμους της Ισπανίας. Να το ξέρουμε αυτό γιατί είναι ευρωπαϊκό το πρόβλημα. Γι' αυτό και πρέπει να το συζητήσουμε και να επιστήσουμε την προσοχή όλων ότι υπάρχει μία εκκρεμότητα. Αυτά είχα να πω. Και τελειώνω ευχαριστώντας την δίκηση της Επιτροπής μας που κατάλαβε ότι το θέμα αυτό, που μπορεί να μην είναι έτσι αυστηρά σαν τα θέματα που εξετάζει η Επιτροπή μας, παρόλα αυτά έχει θέση εδώ στην Επιτροπή αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ και πάνω απ' όλα ευχαριστώ πολύ την κόρη και την εγγονή του Ανσέλμο. Κοιτάξτε τα χαρτιά που έχουμε, τα έγγραφα που έχουμε, είναι, είναι φοβερό. Ο άνθρωπος αυτός σε ένα έγγραφο από ένα Δήμο που έχουμε εδώ στα χέρια μας, που λέει ότι είναι σύνταγματικό μάλιστα Δήμος, έτσι, μιλάει για το Σύνταγμα, τι λέει, λέει ότι πρόκειται για ένα άτομο προωθημένων ιδεών, έτσι το χαρακτηρίζει, ε? αυτό είναι το έγκλημα, προωθημένων ιδεών, επικεφαλής και μασόνου. Έτσι λέει. Είναι, είναι, τρομερά αυτά που διαβάζουμε εδώ. Το άτομο αυτό το οποίο δολοφονήθηκε το 1936, το 43 χαρακτηρίζεται έτσι, Έπτα χρόνια δηλαδή μετά τη δολοφονία, λέει ότι μπορούν να του δοθούν τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία του κατασχέθηκαν τρία χρόνια μετά τη δολοφονία. Κάποια μέρα θα έπρεπε να μελετηθεί και να διαβάσουμε για το πραγματικό ολοκαύτωμα που είχαμε στην Ισπανία μετά τη λήξη του εμφυλίου πολέμου. Προσέξτε, μετά τη λήξη του εμφυλίου πολέμου, όχι κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου και κυρίως αφού θριάβευσε το φασιστικό πραξικόπημα, δεν υπήρξε θέμα εκδίκησης, όχι. Επιστημονικά προετοιμάστηκε το ολοκαύτωμα να εξαφανίσει όλα όσα δεν ταιριάζανε με το ολοκληρωτικό καθεστώς, ακόμα και με την ολοκληρωτική εκκλησία που είχαμε εκείνη την εποχή. Αυτά πρέπει να μελετηθούν ακόμα για να καθαρίσει ο τόπος, που δεν έχει καθαρίσει ακόμα 40 χρόνια μετά. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε με τέτοια υπομονή. Η αλήθεια είναι ότι ναι, δυσκολεύομαι να ολοκληρώσω. Αν δεν σας τα έλεγα αυτά δεν θα ησύχαζα. Σας ευχαριστώ κυρία Ούκεν για 30 δευτερόλεπτα. Θα είμαι πολύ σύντομη. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τον συνάδελφο γιατί διάβασα για το ζήτημα αυτό στις εφημερίδες της Δανίας για τον δικαστή Καρζόν. Ήμουν έξαλλη για αυτό το θέμα. Και ακούγοντα μετά τα παράλογα πράγματα που μας έλεγε η Κομισιόν, δεν μπόρεσα να συγκρατηθώ. Αλλά χαίρομαι για το ότι θα βοηθήσετε για να αποκαλυφθεί η αλήθεια. πρέπει, πρέπει να προσκαλέσουμε τον Παλταζάρ Γκαρθόν εδώ πέρα, να έρθει εδώ και να μας, να μας πει κάποια πράγματα. Γιατί θέλουμε προφανώς να μάθουμε όλοι περισσότερα πράγματα γι' αυτό. Και ήταν καλή ιδέα να, να δώσουμε συνέχεια. Ε, τι να πω, οι προκαταλήψεις μου υπερίσχυσαν. Ένα, ένα λεπτό για, να απαντήσετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Θέλω να κάνω μια διευκρίνηση. Πρώτα απ' όλα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να σας πω ότι εγώ δεν είμαι ούτε δικηγόρος ούτε δική στις ε, οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ό,τι λέτε το δέχομαι. Απλώς διάβασα το χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων σημείο 8.2 που λέει ότι τα δεδομένα προσωπικών δεδομένων εξετάζονται για συγκεκριμένους λόγους και για το άτομο το οποίο είναι το ενδιαφερόμενο ή οποιοδήποτε άλλο που έχει λόγο να ζητήσει, που το αφορούν δηλαδή. Μιλάει για άτομα που τα αφορούν. Άρα δεν πρόκειται μόνο για τα άτομα τα ίδια τα ενδιαφερόμενα, αλλά και για τα άτομα τα οποία αφορούν τα προσωπικά δεδομένα του ατόμου που ζητάει. Μιλάει για θεμητό αίτημα μιλάει για στοιχεία που αφορούν το άτομο, ε? που αφορούν. Δεν είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Άρα δεν είναι πέρα από αυτά που ζητάμε, αλλά επαναλαμβάνω, εγώ δεν είμαι ειδική ούτε δικηγόρος, απλώς διαβάζω. Επίσης θέλω να απαντήσω στον κύριο Ντουράη το εξή. Δεν ήξερα ότι ήταν ε, τόσο σημαντική η αναφορά αυτή και ότι μπορούσε να ανοίξει και την πόρτα στους κράτες και τους Τούρκους, λέει η ομιλήτρια. Είναι ένα θέμα που φαίνεται ανοίγει την πόρτα τόσο το καλύτερο. Αν έτσι βγει κάτι καλό. Για τις ε, διευκρινήσεις όσον αφορά το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ναι. Ψάξαμε σε πάρα πολλά αρχεία των θυμάτων του εμφυλίου πολέμου και της γατορίας για παράδειγμα μας έστειλε μια επιστολή οπότε θέλετε είναι στη διάθεσή σας εκεί ένας υπάλληλο του Υπουργείου Δικαιοσύνης λέει ότι ήρθε σε επαφή με τη φυλακή της Κόρδοβα για παράδειγμα και ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για την παραμονή του εκεί δεν είπα ότι όλα τα αρχεία μας έκλεισαν την πόρτα, όχι αλλά πουθενά δεν λέει στην επιστολή αυτή ότι ήρθαν σε επαφή με την δικαιοσύνη της ε, Κόρτοβα ή της ε, Ποσάδας. Λέει ότι ήρθαν σε επαφή με το Δήμο της Κόρδοβας και με τα... το Λιξερχείο. Είναι πολύ δύσκολο να απευθυνθεί, όπως λέτε και εσείς, σε κάποιο δικαστή. Δεν μπορούμε να πούμε σε ένα δικαστή, μα διαβάστε 70 χρόνια η κυρία ψάχνει να βρει τον πατέρα της. Όχι. Η επιστολή αυτή λοιπόν δεν λέει ποτέ ότι ήρθαν σε επαφή με δικαστές. Με το Δήμο ναι, αλλά με τους δικαστές όχι. Και αυτό θέλω να το υπογραμμίσω, γιατί στην επιστολή αυτή δεν αναφέρεται πουθενά τέτοια επαφή με δικαστές. Η ιδέα αυτή να σταλεί η επιστολή στο Δήμο, ναι, αλλά ο Δήμος δεν έχει, έχει μόνο πολιτιστικά αρχεία, δεν έχει δεδομένα. Ίσως, όπως λέτε εσείς, να έχουν καταστραφεί. Ίσως να τα φάγαν τα ποντίκια από το 43 μέχρι σήμερα. Αλλά στο το ψάξουν. Ας το ψάξουν. Ε, λίγο χρόνο χρειάζεται. Εγώ προσωπικά θα πήγαινα, τους λείπει προσωπικό, να πάω εγώ να ψάξω στο Ποσάδας, αλλά να μου ανοίξουν την πόρτα τουλάχιστον. Αυτό σας ζητάω. Εμένα δεν μου απάντησαν, μου απάντησαν διάφορα αρχεία. Αλλά αυτό το συγκεκριμένο όχι, ούτε τηλέφωνο δεν με πήραν. Δεν ξέρω για το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Εντάξει, εσεί. τώρα που κυβερνάτε, αν μπορείτε να έρθετε σε επαφή με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το καλύτερο. Κύριε Τουργάς, 30 δευτερόλεπτα, έτσι. Ναι, ναι, πολύ σύντομα. Για το Υπουργείο Δικαιοσύνη. Σα είπα ότι μου είπαν ότι ήρθαν σε επαφή με δικαστέ από το Ποσάδας και την Κόρδοβα. Και εσείς μιλάτε με το Υπουργείο Δικαιοσύνη. Εγώ να σας πω ποιος είναι να σας δώσω το όνομα και να έρθετε σε επαφή μαζί του. Μπορεί να είναι λάθος. Ε, εντάξει, θα το μάθετε. Όμως, μιλήσατε για τους Κουράτες και για τους Τούρκους. Όχι, όχι. Είναι οι Κύπροι μετά την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο. Υπάρχουν πάρα πολλοί αγνοούμενοι και πάρα πολλές μανάδες που ψάχνουν τα παιδιά τους ε, από την Κύπρο. Οι Κύπριώτες οι Κύπροι λοιπόν, οι Κροάτες κλπ. Όντως, αλλά εκτό από αυτού υπάρχουν τις κι εκατομμύρια Ευρωπαίοι, παιδιά, γυναίκες, εγγόνια που ψάχνουν τους αγνούμενου τους. Και γι' αυτό λέω ότι και εγώ θα ήθελα πάρα πολύ όλοι αυτοί οι άνθρωποι να βρούνε κάποια λύση στο δράμα τους και να μάθουν τι έχει γίνει με τους δικούς τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ που ήρθατε και κάναμε αυτή την πολύ έντονη συζήτηση και εις βάθος συζήτηση. Νομίζω πως είμαστε όλοι σύμφωνοι πέρα από κάποιους ε, προγραμματισμούς κάπως διαφορετικού. Τα πορίσματά μας ε, πρέπει να είναι κοινά και ομόφωνα. Να αφήσουμε ανοιχτό το αίτημα, την αναφορά. ως επίπτωση της αρμοδιότητας μας να κάνουμε μια έκκληση στις Ισπανικές Αρχές, στον Υπουργό Δικαιοσύνης της Ισπανίας συγκεκριμένα, για να τον καλέσουμε, να του θυμίσουμε ε, αυτά που θα έπρεπε να είναι τα καθήκοντα μιας ε, δημοκρατικής ε, εξουσίας, να προσθέσουμε ένα συμπλήρωμα νέο στην Εκτελεστική Επιτροπή για να γνωστοποιήσουμε στην ίδια την Επιτροπή ότι επί τη βάση των επιχειρημάτων που εκφράσατε θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει μια παραπάνω προσπάθεια αναλυτική για να επαληθεύσουμε και να εφαρμόσουμε πλήρως την αρχή της επικουρικότητας που είναι βασική στη, στα θεσμικά μας όργανα και που σίγουρα δίνει στο θεσμικό όργανο που είναι πιο κοντά στον πολίτη το καθήκον και το δικαίωμα να ασχοληθεί όπως λέει και η Κομισιόν στο σημείο τη, αλλά σε περίπτωση καταλληλότητας η αρχή αυτή λέει ότι μπορούμε να φτάσουμε ακόμα και στα θεσμικά όργανα για την προστασία των δικαιωμάτων όταν ε, τα θεσμικά όργανα που είναι πιο κοντά στον ίδιο τον πολίτη δεν το κάνουν. Άρα λοιπόν στο πλαίσιο των θεμελιωδών δικαιωμάτων αντίθετα με τα όσα λέει η Κομισιόν υποστηρίζει Κομισιόν υπάρχει αρμοδιότητα των ε, ευρωπαϊκών θεσμών, δηλαδή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί συνεχίζεται η παραβίαση κάποιων από αυτά τα δικαιώματα, όπως ε, προέκυψε από αυτήν εδώ την υπόθεση. Έπειτα, σε σχέση με την αδυναμία παρέμβασης εκεί όπου πρόκειται για πληροφορίες που αφορούν τρίτους. Αυτή η ερμηνεία είναι κάπως περιοριστική και θα πρέπει να σας πω ότι η Επιτροπή έδωσε με βάση μάλλον την οδηγία περί δικαιώματος ενημέρωσης των πολιτών, νομίζω προέκυψε κοινή βούληση να ζητήσουμε μια, ένα, μια περαιτέρω εμβάθυνση από την Κομισιόν. Σας ευχαριστώ πολύ κυρίες μου λοιπόν που ήρθατε και που πήρατε το λόγο εδώ. Μια ακόμη πρόταση, ναι. Κυρία Πρόεδρε, εγώ συμφωνώ απόλυτα με την πρότασή σας, αλλά μετά από την παρέμβαση του κυρίου Τουργκάης και εγώ θα ήθελα να σας ε, πω ότι στην τοπική ε, κυβέρνηση της Ανδαλουσίας ε, εγώ και ο συνάδελφος είμαστε στην κυβέρνηση, σε κόμματα που είναι στην κυβέρνηση και νομίζω ότι θα πρέπει να τεθεί το θέμα και να εξυπηρετήσουμε με τους αρμόδιους της κυβέρνησης της Ανδελουσίας ε, το συγκεκριμένο θέμα. Σας ευχαριστώ που μου το είπατε. Αν δεν είχατε καταλάβει την παρέμβασή μου, είπα για εθνικές τοπικές αρχές, όπως πρότεινε και ο κύριος Μαρτίνες Μαρτίνες στην δική του παρέμβαση. Δηλαδή θα στραφούμε και στους δύο άμεσα ως Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ και πάλι και αφήνω την Προεδρία στον συνάδελφο Μέγερ. voy a despedirme de voy a, voy a despedirme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 Συνεχίζουμε παρακαλώ. Τα πηγαδάκια εκτός αιθούσης παρακαλώ. Γιατί υπάρχει και επόμενη αναφορά και νομίζω ότι οι αναφέροντες είναι εδώ, έτσι. Πρόκειται για την αναφορά 791 καθέτος 2008 του Κρίστοφερ Στόκουελ, Βρετανικής Ιθαγένεια, εξ ονόματο. 15. Ναι. Α, όχι, στη 16 πάμε. Αναφορά 1032-2010 του Μανουέλ Αλτεμίρ Μερχελίνε, Ισπανική Στεγέννη, σχετικά με τη διακριτική μεταχείριση που υφίσταται οι μαθητέ των Ευρωπαϊκών Σχολείων κατά την πρόσβασή του στα Ισπανικά Πανεπιστήμια. Το λόγο έχει ο κύριο Μανουέλ Αλτεμίρ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τουργαϊδ. Πρώτα απ' όλα να δηλώσω και εγώ τη στήριξή μου στην οικογένεια που είχε την προηγούμενη αναφορά και να πω ότι τους θαυμάζω για το θάρρος τους για ένα τόσο δύσκολο θέμα. Τώρα εγώ ήρθα εδώ σήμερα για να σας μιλήσω για ένα θέμα λιγότερο σημαντικό. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο αυτό, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν είναι και πρόβλημα παρόλα αυτά. Και το πρόβλημα είναι μια αδικία που πιστεύω ότι γίνεται σε βάρος των μαθητών των ευρωπαϊκών σχολείων και άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν αυτοί θέλουν να μπουν στο Πανεπιστήμιο το Ισπανικό, στην Ισπανία. Οι μαθητές ε, αυτοί αντιμετωπίζουν δυσκολία για να μπουν στα Ισπανικά Πανεπιστήμια. Αυτό είναι αδιαφυσβήτητο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρεται στις δυσκολίες αυτές η ίδια στην ανακοίνωσή της που έχει η Επιτροπή σας. Υπάρχουν στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι οι Ισπανοί μαθητές των ευρωπαϊκών σχολείων είναι εκείνοι οι οποίοι πάνε λιγότερο από όλους τους άλλους στα Ισπανικά πανεπιστήμια. Υπάρχει το παράρτημα 5 της ε, μελέτες που ζητήσατε εσείς ήδη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και που έχει ως τίτλο Analysis of the Academic and Professional Careers of the European Schools Graduates του Οκτωβρίου του 2008 όπου οι συντάκτες της μελέτης αυτής καταδεικνύουν ότι ενώ είναι 70% περίπου οι μαθητές από τις ε, άλλες χώρες επιστρέφουν στις χώρες τους για να σπουδάσουν. Ε, λοιπόν, όσον αφορά τους Ισπανούς, μόνο το 51% μπαίνει στα Ισπανικά πανεπιστήμια. Επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ανακοίνωση που έστειλε στην ε, Επιτροπή σας αναφέρεται σε μια ομάδα εργασίας που δημιουργήθηκε προκειμένου να επιτευχθεί μια λύση στο πρόβλημα αυτό. Δηλαδή σημαίνει ότι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές του Ισπανικού τμήματος υπάρχουν. Είναι αδιαφεσβήτητες. Τώρα, ποια είναι η πηγή του προβλήματος. Το πρόβλημα είναι εξαιτία των ε, ισπανικών προδιαγραφών που μειώνουν τους βαθμούς που έχουν πάρει οι Ισπανοί μαθητές των ευρωπαϊκών ε, σχολείων ε, σε σύγκριση με τους υπόλοιπους. Και γιατί, γιατί στην Ισπανία για να περάσει κανείς χρειάζεται να πάρει 5 στα 10 βαθμό. Στα ευρωπαϊκά σχολεία όμως και σε άλλα, ενδεχομένω είναι πιο ποτητική και δεν ε, θέλουν 5 στα 10, θέλουν 6 στα 10 για να προβιβαστεί κανείς. Και τι κάνουν λοιπόν οι Ισπανοί? Λένε ότι το 6 που παίρνει ένας μαθητής του Ευρωπαϊκού Σχολείου είναι το ίδιο όπως ένα 5 που παίρνει ένας μαθητής στα Ισπανικά σχολεία. Αυτό είναι παράδοξο για μένα. Γιατί παρόλο που χρειάζονται παραπάνω απαιτήσει από τα ευρωπαϊκά σχολεία για να περάσει κανείς, ε, παρόλα αυτά ζημιώνονται σε σύγκριση με τους Ισπανούς μαθητές και έτσι δυσκολεύονται πιο πολύ να μπουν στο πανεπιστήμιο της χώρας τους. Και μιλάω για τους μαθητές των Ευρωπαϊκών Σχολείων και ιδιαίτερα του Ισπανικού τμήματος, γιατί εκεί έχω και εγώ τα παιδιά μου. Το πρόβλημα αυτό όμως δεν αφορά μόνο αυτούς, έχει να κάνει και με τους άλλους μαθητές των Ευρωπαϊκών ε, Σχολείων αν ε, ένας Γάλλος μαθητής θέλει να πάει σε Ισπανικό Πανεπιστήμιο, πάλι το ίδιο πρόβλημα θα έχει. Το ίδιο ισχύει και με ε, μαθητές από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θέλουν να πάνε να σπουδάσουν στην Ισπανία. Αυτές οι ισπανικές προδιαγραφές λοιπόν αντιβαίνουν στην αρχή της ελεύθερη κυκλοφορία των ατόμων και των εργαζομένων, αρχέ οι οποίες ε, καθορίζονται από τι συνθήκες. παραβιάζουν επίσης και άλλες ευρωπαϊκές προδιαγραφές όπως είναι η Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και το άρθρο 5 της Διακυβερνητικής Σύμβασης που αναφέρεται στο καθεστώς των Ευρωπαϊκών Σχολείων. Ποια είναι η άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πριν έρθουμε εδώ, ε, υποβάλαμε προσφυγή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε τρία σημεία συνοψίστη απάντηση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρώτον, λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι οι χώρε μέλη είναι οι μόνε επέθυνοι... για την οργάνωση των εκπαιδευτικών συστημάτων του. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό. Λέει επίση ότι οι προδιαγραφέ αυτέ δεν θα πρέπει να δυσκολεύουν τους μαθητές με απολυτήριο από άλλο σχολείο. Και εδώ συμφωνώ. Όμως, πιστεύω ότι οι ισπανικές ε, προδιαγραφές ζημιώνουν και χωρίς λόγο τους ε, μαθητές από άλλα σχολεία. Λέει επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν υπάρχει προφανής παραβίαση του ευρωπαϊκού δικαίου. Δεν συμφωνώ όμως. Εγώ καταλαβαίνω ότι οι ισπανικές προδιαγραφές αυτό που προσπαθούν να κάνουν είναι να πετύχουν ότι όλοι οι μαθητές βρίσκονται στην ίδια κατάσταση τη στιγμή που μπαίνουν στο Ισπανικό Πανεπιστήμιο. Όμως είναι πολύ σημαντικό η βαθμολογία που έχει κανείς από το πολιτήριό του, γιατί ανάλογα με τη βαθμολογία αυτή μπορεί να μπει στη μία ή την άλλη σχολή του Ισπανικού Πανεπιστημίου, γιατί απαιτούνται υψηλέ βαθμολογίε μερικέ φορέ για να μπει κανεί στη σχολή που θέλει. Οι Ισπανικέ αρχέ λοιπόν δεν μπορούν να λένε ότι πετυχαίνουν την ε, ισοτιμία. Κάνουν ακριβώ το αντίθετο. Ζημιώνουν αδικαιολόγητα ορισμένους μαθητές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει επίσης ότι οι Ισπανικές Αρχές δεν πρέπει να λάβουν υπόψη τους ε, το, τις απαιτήσει άλλων εκπαιδευτικών ε, συστημάτων όταν κάνει την μετατροπή. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό. Δεν συμφωνώ με αυτό. Μπορώ να συμφωνήσω εφόσον οι ισπανικές προδιαγραφές δεν κάνουν καμία μετατροπή. Αλλά από τη στιγμή που μειώνουν τη βαθμολογία, θα έπρεπε να έχει γίνει κάποια μελέτη για να δούμε κατά πόσο δικαιολογείται ή όχι αυτή η μετατροπή, αυτή η μείωση δηλαδή. Πράγμα το οποίο δεν έχει γίνει στην Ισπανία. Γι' αυτό για μένα η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην αναφορά μου είναι πολύ απλουστευτική και ξεκινάει από λάθος βάση. Τώρα γιατί εισήγαγα την, ε, υπέβαλα μάλλον την αναφορά αυτή στην Επιτροπή σας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρώτα όλα, επειδή οι προσπάθειες που έχω κάνει μέχρι τώρα για να βρω μια λύση σε φιλικό επίπεδο με τις ε, μέχρι τώρα ισπανικές κυβερνήσεις δεν απέφερε καρπούς. Παρά τις ε, συνεχείς προσπάθειες των οργανώσεων των ε, γονέων των μαθητών και τις επαναλημμένες επιστολές που έχουμε στείλει στον Επίτροπο Κάλλας. Τίποτα δεν έγινε. Περνάει ο χρόνος, τα παιδιά μου μεγαλώνουν, όπου να είναι θα πρέπει να πάνε στο πανεπιστήμιο και δεν υπάρχει λύση υπήρξε αλλαγή στην κυβέρνηση στην Ισπανία, πράγματι. Το καλύτερο, ο καλύτερος τρόπος για να βρεθεί λύση είναι με έναν φιλικό διακανονισμό. Οποιαδήποτε λοιπόν αλλαγή στη στάση των Ισπανικών αρχών είναι ευπρόσδεκτη. Τώρα, ε, επαγγελματικά, εγώ είμαι υπάλληλο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γνωρίζω ότι το να απευθυνθεί κάνει στην Επιτροπή σας είναι πολύ χρήσιμο. Είναι επίσης πολύ χρήσιμο να υπάρχουν προσφυγές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ προσωπικά δουλεύω στην ε, Γενική Διεύθυνση για την Φορολογία και τα Τελωνία. Έξι χρόνια τώρα. Στην ε, Μονάδα για τις Παραβιάσεις. Πρέπει να σας πω λοιπόν ότι τα τελευταία δέκα χρόνια έχω διαπιστώσει ότι εθνικές πρακτικές και προδιαγραφές που θεωρώντουσαν ιερές μετά από δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν ισχύουν πια. Έτσι έχουν καταργηθεί εμπόδια που αντιμετώπιζαν οι Ευρωπαίοι πολίτες προκειμένου να κυκλοφορήσουν ελεύθερα στον ευρωπαϊκό χώρο. Υπάρχει επίσης και αυτή η μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2011 στα αγγλικά. Ο τίτλος είναι the impact of the rulings European Court of Justice in the area of direct taxation 2010. Είναι 200 σελίδες περίπου όπου σχολιάζονται οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για θέματα άμεσης φορολόγησης. Υπάρχουν μερικέ γενικέ διευθύνσει λοιπόν μέσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που δραστηριοποιούνται περισσότερο από άλλε προκειμένου να θέσουν υπομφισβήτηση εθνικές προδιαγραφές. Δεν έχω βέβαια μεγάλη εμπειρία για να μπορώ να πω τι κάνει η Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θεωρώ όμως ότι μια τέτοια προσφυγή στην Γενική Διεύθυνση θα έπρεπε να έχει λάβει κάποια μεγαλύτερη προσοχή και συνέχεια. Θέλω επίσης να αναφερθώ εδώ και σε έναν ανακοινωθέν τύπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του, της 26 Οκτωβρίου πριν μερικές εβδομάδες δηλαδή όπου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητάει την άρση των εμποδίων στην εσωτερική καινή αγορά. Και εκεί αναφέρονται διάφορα θέματα που είναι σε κρεμότητα, όπως είναι τα τέλη κυκλοφορίας των ε, οχημάτων όταν ε, φεύγουν από μια χώρα και πηγαίνουν σε μια άλλη, ε, οι δυσκολίες προκειμένου να ανοίξει κανείς τρέχοντα λογαριασμό στην τράπεζα. Αλλά υπάρχει και αυτό το πρόβλημα που σα αναφέρω εγώ. Εγώ δεν θα ήθελα τα παιδιά μου να πληρώσουν την ύφη επειδή εγώ αποφάσισα να έρθω να δουλέψω εδώ στι Βρυξέλλες και τα παιδιά μου πάνε στο Ευρωπαϊκό Σχολείο. Δεν θα ήθελα μια τέτοια διάταξη που πιστεύω ότι είναι άδικη και τα τιμωρία δίκως να συνεχίσει να ισχύει. Σα ζητάω να κοιτάξετε το θέμα, να το αναλύσετε από νομική άποψη. Είμαι στη διάθεσή σας απόλυτα προκειμένου να σας δώσω ό,τι πληροφορίες έχω στα χέρια μου και σας ζητάω παρακαλώ να κάνετε ό,τι περνάει από το χέρι σας για να αλλάξει η ισπανική νομοθεσία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Δον Μανουέλ. Άμα ξέρετε την Επιτροπή των Αναφορών, ξέρετε ότι τώρα θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να απαντήσει. Και θα απαντήσει ο κύριος Βάλτερ Τσαμπίν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ να ξεκαθαρίσω την νομική πτυχή και μετά θα δώσω τον λόγο στο συνάδελφο και θα εξηγήσω στον συνάδελφο στο διάλογο που έχουμε με τις Ισπανικές αρχές. Όπως βλέπετε ο αναφέρον έχει ήδη κάνει μια σύνοψη. Εμείς συμφωνούμε θεμελιωδώς. Θεωρούμε πως οι Ισπανικές αρχές είναι εντός των αρμοδιοτήτων τους όταν κάνουν μετατροπή τη βαθμολογίας του Ευρωπαϊκού Σχολείου στο δικό τους σύστημα. Βεβαίω, ε, επειδή και οι δύο κλίμακες βαθμολογίες είναι στο 10 ε, κάνει το επιχείρημα σε μια πρώτη ανάγνωση να φαίνεται λογικό. Αν ήταν ε δεν θα το συζητούσαμε. Αλλά σημασία έχει ποια είναι η βάση. Συγκρίνουν λοιπόν οι Ισπανικές αρχές μια βάση 6 βαθμών πάνω από τη βάση με μια που είναι 5 ε, που έχει 5 βαθμούς πάνω από τη βάση που είναι η Ευρωπαϊκή. Εμείς δεν θεωρούμε πως υπάρχει κάποια παράβαση. Δεν βλέπουμε πως υπάρχει εδώ πέρα παράβαση. Για να είμαι ξεκάθαρος για τον συνάδελφο. Στον τομέα της εσωτερική αγοράς αρκεί να αποδείξουμε πως υπάρχει φραγμός. Στον τομέα της εκπαίδευσης όμως πρέπει να αποδείξουμε διάκριση που είναι κάτι το πολύ πιο δύσκολο να αποδειχθεί. δεν ξέρω ειλικρινά τι άλλο να προσθέσω. Νόμιζα πως είχαμε ήδη εξηγήσει τη θέση μας γραπτός και σε επανειλημμένη επικοινωνία που είχαμε με τον αναφέροντα πριν. Γιατί είχαμε στείλει αυτή την απάντηση. Σας ευχαριστώ. Η συνάδελφό σας έχει τον λόγο. Είμαι η Μαρή Σέντερ από τη Γενική Διεύθυνση Προσωπικού για, υπεύθυνη για τα ευρωπαϊκά σχολεία. Να πω κάποια πράγματα. Είναι συνεχές το πρόβλημα ε, σε όλα τα κράτη-μέλη να γίνει η μετατροπή του μπακαλωρεά ε, με το σύστημα του κάθε μέλους. Οι επιθεωρητές που έρχονται από τα Υπουργεία Παιδείας, στα εθνικά, ξέρουν το σύστημά τους καλύτερα. Και η Κομισιόν έχει έρθει σε επαφή με τους Ισπανούς επιθεωρητές για να αντιληφθεί τη, τη λογική τους και όπως εξήγησε ο συνάδελφος, η αξιολόγηση την οποία κάνουν βασίζεται στη δική τους πείρα. Το σύστημα του Ευρωπαϊκού Σχολείου αυτή τη στιγμή τι γίνεται. Υπάρχει ε, μια τεχνική ομάδα εργασίας αρμόδια για το Ευρωπαϊκό Μπακαλωρεά που αξιολογεί την κλίμακα βαθμολογίας για να γίνει πιο διαφανής αυτή για να μπορέσουν τα κράτη-μέλη να κάνουν την μετατροπή. Ε, είναι ένα έργο εν αλλάζει η διδακτέα ύλη συνεχώς και είναι πράγματα τα οποία παρακολουθούμε και μπορούμε νομίζω έτσι να κάνουμε το σύστημά μας ε, πιο διαφανές ε, για να μπορεί να γίνει αυτή η, η αξιολόγηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Θέλει κάποιος άλλος το λόγο πριν ε, ο αναφέρον ε, απαντήσει. Θέλετε να απαντήσετε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εντάξει, έχετε το λόγο. Ναι, θέλω να διευκρινίσω κάτι, να μην πω βέβαια σε λεπτομέρειες, αλλά βλέπω κάθε εβδομάδα τι γίνεται με τις εξετάσεις των ε, παιδιών μου. Αν έχουν 10 ερωτήσεις και απαντήσουν στις 5, κόβονται. Αν απαντήσουν στις 6, περνάνε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει, και το λένε και κάποια έγγραφα, ότι το γεγονός ότι στα ευρωπαϊκά σχολεία χρειάζεσαι έξι για να περάσεις, αυτό επηρεάζει και τη βαθμολογία που δίνει ο καθηγητής. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι λάθος. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Η κατάσταση είναι ξεκάθαρη και για μένα Προφανώς και υπάρχει διάκριση. Αν βάλω το γιο μου να δώσει εξετάσεις και πάρει έξι και βάλω τον ξάδερφό του που είναι στη Μαδρίτη και πάρει πέντε, όταν φτάσουν για να μπουν στο πανεπιστήμιο και οι δύο θα έχουν πέντε. Έχω έξι χρόνια που δουλεύω πάνω σε αυτά τα θέματα, όχι βέβαια στην εκπαίδευση και στον πολιτισμό, δεν ξέρω τη διαφορά ανάμεσα στη διάκριση και το εμπόδιο. Εγώ βλέπω ότι υπάρχει μια διάκριση και ότι δεν αιτιολογείται η ρύθμιση αυτή που έχουν οι Ισπανικές αρχές. Εγώ πιστεύω ότι ζημιώνονται τα δικά μου τα παιδιά και θέλω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει κάτι παραπάνω και θεωρώ ότι μπορεί. Δεν καταλαβαίνω τη θέση της. Πιστεύω ότι σε περίπτωση αμφιβολίας πάμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για να αποφανθεί εκείνο. Αυτό ζητάω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κοιτάξτε το θέμα με τη νομική σας υπηρεσία. Αν θεωρείτε ότι πρέπει να με υποστηρίξετε, πιέστε την Επιτροπή ή κάντε ό,τι νομίζετε. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι πρόκειται για διάκριση και τα επιχειρήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν με πείθουν. Όσο και αυτά που είπε η εκπρόσωπος ε, των ανθρώπινων πόρων. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ, αλλά εγώ σας το είπα και πριν, περνάει ο χρόνος. Το να δημιουργούνται ομάδες εργασίας που να δουλεύουν με διαφάνεια και τα λοιπά Πολύ ωραία, αλλά έχουν περάσει τόσα χρόνια. Και κάθε χρόνο υπάρχουν τουλάχιστον 50 Ισπανοί μαθητές οι οποίοι ζημιώνονται από αυτό το θέμα. Και μιλάμε για ανθρώπους έτσι, μιλάμε για παιδιά 17 χρονών το καταλάβατε. Δεν μπορούν δηλαδή επίσης όρις να αποφασίσουν πού θα σπουδάσουν. Για μένα αυτό είναι αδικία. Ευχαριστούμε πολύ, Δον Μανουέλ. Σας αντιλαμβάνομαι, καταλαβαίνω. Πιστεύω και εγώ ότι υπάρχει μια διάκριση εδώ. Πολύ καλά μας τα εξηγήσατε όλα. Επιτρέψτε μου τώρα μια που θα παραμείνει ανοιχτή η αναφορά, γιατί εγώ ζητάω να μείνει ανοιχτή. Και έτσι γίνεται. Αν υπάρχει ένας βουλευτής που ζητάει να μείνει ανοιχτή μια αναφορά, μένει ανοιχτή. Επιπλέον, γιατί και η Επιτροπή δείχνει να υπάρχουν αμφιβολίες για αυτό το θέμα. Συνεπώς, αν συμφωνείτε, θα στείλουμε επιστολή στο Διευθυντή των Ευρωπαϊκών Σχολείων να το εξηγήσουμε αυτό το θέμα και να του ζητήσουμε τη γνώμη του. Οι νομικές υπηρεσίε δεν ξέρω. Εννοούσατε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή τις δικέ μα νομικές υπηρεσίε εννοούσατε. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Και δεν ξέρω αν θέλετε η Ισπανική κυβέρνηση να πει κάτι, γιατί θα μπορούσαμε να ζητήσουμε από την Ισπανική κυβέρνηση να μα πει. Εσεί θα έχετε πάρει επαφή με την Ισπανική κυβέρνηση, έτσι δεν είναι. Τα τελευταία νέα που έχω είναι ότι, ότι υπήρξε επαφή με την προηγούμενη κυβέρνηση. Με αυτή την κυβέρνηση δεν ξέρω. Ωραία, τότε να το κάνουμε και αυτό. Να στείλουμε μια επιστολή στο Υπουργείο Παιδείας. Η γραμματεία να το σημειώσει. Μένει ανοιχτή λοιπόν αυτή η αναφορά, περιμένοντας τι απάντηση θα πάρουμε και ανάλογα θα δούμε τι συνέχεια θα δώσουμε. Ευχαριστούμε τον Μανουέλ. Αναφορά 17 του 1997 καθώ 2011 Το Άλμπερτ Φαντεχάν, Ολλανδική Ιθαγένεια Ξενόμητο Ομοσπονδία Ευρωπαίων Δημοσίων Λειτουργών, FFPE, η οποία συνοδεύεται από περίπου 60 υπογραφέ σχετικά με τη χορήγηση εκπαιδευτικού επιδόματο σε προσωπικό του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλώματων Εύρεση Τεχνία. Ο κύριο Άλτερ Γιάν Τεχάν είναι εδώ, έτσι δεν είναι. Dear Αγαπητά μέλη της Επιτροπής, σας ευχαριστώ που με επιτρέπετε να παρουσιάσω την αναφορή μου. Λέγομαι Άλτερ Τιάντε Χάν, Ολλανδός υπήκος και υπάλληλο του Ευρωπαϊκού Γραφείου Ευρεστεχνία στην Ολλανδία. Αυτή τη στιγμή δεν εκπροσωπώ την υπηρεσία μου, αλλά το συνδικάτο FFP και τους 63 συναδέλφους που υπέγραψαν αυτή την αναφορά. Το πρωτοδικείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε το 2003 πως είναι παράνομο να συνδέεται το επίδομα εκπατρισμού με το επίδομα εκπαίδευσης και υπάρχει κανόνα στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης που απαγορεύει να αποσυνδέεται να συνδέεται, με συγχωρείτε, να συνδέονται τα δύο επιδόματα. Αυτό επηρεάζει βεβαίως τους Αυστριακούς ε, στην Βιέννη, τους Γερμανούς στη Γερμανία και τους Ολλανδούς ε, στη Χάγη, όλους στην ίδια υπηρεσία. Ε, διαμαρτυρόμαστε εδώ και πάρα πολλά χρόνια για αυτή τη διάκριση με βάση την εθνικότητα και θεωρούμε πως πρόκειται για παραβίαση του άρθρου 21 της Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Έχουμε υποβάλει επίσης προσφυγή στην Γενέβη στο δικαστήριο του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας το οποίο δεν ε, εφάρμοσε την ομολογία του ε, ΔΕΚ και η υπηρεσία μας η ίδια θεώρησε ότι δεν δεσμεύεται από την ομολογία του ΔΕΚ. Η ανάλυση της Κομισιόν εδώ πέρα δεν είναι πλήρης. Η Κομισιόν παραδέχεται πως όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι επίσης ε, κράτη-μέλη του Ευρωπαϊκού Γραφείου ε, του διπλωμάτων ευρεσιτεχνία. Η υπόθεση 8C8 του 2008 ξεκαθάρισε πώ οι εκπρόσωποι των κρατών μελών είναι υπεύθυνοι για να διασφαλίσουν την τήρηση των κανόνων του κοινοτικού δικαίου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του. Αυτό σημαίνει πω οι 27 εκπρόσωποι των κρατών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Γραφείου Ευρεσιτεχνία πρέπει να φροντίσουν για την τήρηση των αρχών του κοινοτικού δικαίου και του κανονισμού του οργανισμού μας. Επίσης, η Κομισιόν δεν αναφέρει πως η ίδια έχει καθεστώς παρατηρητή στο Διοικητικό Συμβούλιο. Υπάρχει και η περίπτωση C34 κάθετος 10 Crystal κατά Greenpeace στο 10 για την ε, ερμηνεία της οδηγίας για τις βιοτεχνολογικές εφευρέσεις. Θα δεχόταν σε αυτή την περίπτωση πως ε, η υπηρεσία μας δεν δεσμεύεται από την ε, νομολογία και δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Εάν η Κομισιόν δεν είναι αρμόδια για κάτι το οποίο συμβαίνει το, στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνία, όπου συμμετέχουν και τα 27 κρατη μήπω αυτό θα έπρεπε να ανισχύσει λίγο το Κοινοβούλιο θα ήθελα να αφαιρθώ σε μια δήλωση του Ρόκο Μπουτιλιώνη στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 30 Μαρτίου 2000 για το δίπλωμα ευρεσιτεχνία που ζητήθηκε για γενετικά τροπημένα ανθρώπινα έμβρια. Είπε, υπάρχει έλλειμμα στον νόμο. Δεν είναι δυνατόν το Ευρωπαϊκό Γραφείο Ευρεσιτεχνία να μην έχει σχέση και επαφή με την Κομισιόν ή να μην είναι μέρο της δομής Ευρωπαϊκής Ένωσης, κλείνουν τα εισαγωγικά. Γι' αυτό η Κομισιόν δεν μπορεί να δηλώσει αναρμόδια για την κατάσταση στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Ευρεσιτεχνίας. Το πρόβλημα που παρουσιάζουμε εδώ πέρα αφορά Ευρωπαίους πολίτες οι οποίοι εργάζονται σε μια υπηρεσία που όλες τις υπηρεσίες βρίσκονται στο Μόναχο, Βερολίνο, Βερολίνο Βιέννη και Χάγη, δηλαδή εντός της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά τώρα την παρέμβαση που ζητάμε από το Κοινοβούλιο και την Κομισιόν, θέλουμε να αφαιρθούμε στην παρέμβαση τη Κομισιόν στο ΔΟΥΣΟΥ του οργανισμού μα τον Οκτώβριο του 2004 για το ζήτημα τη ε, αναγνώριση από την υπηρεσία μα σχέσεων του ιδίου φύλου. Η παρέμβαση αυτή τη Κομισιόν που ήταν αποτέλεσμα ερώτηση Ευρωβουλευτού τη κυρία Σόφι Ινετφέλτ έχει δείξει πω είναι δυνατόν η Κομισιόν να παρεμβαίνει για εσωτερικά ζητήματα Τη υπηρεσία. Αυτό το οποίο ζητάμε τώρα είναι η Κομισιόν να παρέμβει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Γραφείου για να υπάρξει συμμόρφωση με την ομολογία του Πορτοδικίου για το επίδομα εκπαίδευση. Συνελώντη λοιπόν. Ζητάμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δώσει οδηγίε στην Κομισιόν να παρέμβει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνία, να υπενθυμίσει δηλαδή στι 27 αντιπροσωπείε των κρατών μελών την υποχρέωσή τους να συμμορφωθούν με την ομολογία του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όσον αφορά το επίδομα εκπαίδευσης και να προσαρμόσουν αναλόγως το άρθρο, 20, το άρθρο 71 του Οργανισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης. Και θα τελειώσω μια ερώτηση. Δέχεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πως ε, είναι δυνατόν να δηλώνει η Ευρωπαϊκή, το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων υπηρεσίες πως δεν δεσμεύεται από την ομολογία του ΔΕΚ. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε, κύριε Γιάνντε Χάν. Θα δώσω λόγο τώρα στον κύριο Λασάλας, ο οποίος θα μιλήσει ξανά της Κομισιόν. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η Κομισιόν εξέτασε λεπτομερώς την αναφορά και αντιλαμβάνεται την θέση του αναφέροντος. Η Κομισιόν λυπάται για το ότι εδώ πέρα δεν μπορεί να συμφωνήσει και μάλιστα για πολλούς λόγους. Πρώτον, όπως έχουμε ήδη πει γραπτός, το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρωστηχνίας είναι άλλο έχει ξεχωριστή νομική προσωπικότητα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μέλος και δεν έχει ψήφο καν στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καθεστώς παρατηρητή και εκπροσωπείται από την Κομισιόν στο Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά, όπως είπα, δεν έχει ψήφο, δεν μπορεί να ψηφίσει. Το ζήτημα λοιπόν εδώ πέρα είναι το εάν πρέπει να αλλάξει το καταστατικό των υπαλλήλων ε, του Ευρωπαϊκού Γραφείου Ευρεσιτεχνίας μετά από μια απόφαση του δικαστηρίου του ΑΕΛΟ. Εμείς θεωρούμε πως πρέπει να τα αποφασίσει αυτά τα ζητήματα το ίδιο το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και η Κομισιόν και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ πέρα δεν θα λάβει γιατί πρόκειται για απόφαση του αρμοδίου δικαστηρίου. Αυτή η απόφαση είναι διαφορετική με την περίπτωση του 2004 την οποία αναφέρατε για τις ε, συμβιώσεις δύο φύλων. Δεν υπήρχε τότε δικαστική απόφαση και η Κομισιόν τότε το 2004 όπως σωστά είπατε ε, τοποθετήθηκε για αυτό το θέμα. Σήμερα όμως η κατάσταση είναι διαφορετική. Υπάρχει μια απόφαση δικαστηρίου. Η Κομισιόν θεωρεί πως επαφίεται στα κράτη-μέλη αν θα αντιδράσουν σε αυτή την απόφαση του δικαστηρίου με μια αλλαγή του καταστατικού ή όχι. Η κατάσταση επίσης διαφέρει και από αυτά τα οποία αναφέρατε για περιπτώσεις ευρεσιτεχνίας. Όταν τοποθετείται εκεί πέρα η Κομισιόν κάτι το οποίο το κάνει τακτικά δεν πρόκειται για εσωτερικές υποθέσεις του οργανισμού αυτού αλλά για ουσιαστικά και εξειδικευμένα ζητήματα δικαίου ευρεσιτεχνίας. Και εκεί πέρα πράγματι τοποθετείται τακτικά η Κομισιόν. Αυτό είναι τελείω διαφορετική φύση ζήτημα από αυτό που μα απασχολεί τώρα. Ευχαριστώ. Ε, Κύριο Γιάρ, ευχαριστώ. Οι νομικέ πληροφορίε που μα έδωσε η Κομισιόν είναι σαφεί εδώ πέρα. Από την άλλη όμω ε, είναι και πολιτικό το ζήτημα. Το εάν δηλαδή θέλουμε να αλλάξουν οι συνθήκες ή όχι. Αυτό το οποίο θα μπορούσαμε να προσφέρουμε στους αναφέροντες, κατά την άποψή μου, είναι να παραπέμψουμε το ζήτημα αυτό στις αρμόδιες επιτροπές για μια γνωμοδότηση, η Επιτροπή δηλαδή Απασχόλησης και η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, αν και... Να μας πούν δηλαδή το εάν επιτρέπονται αυτές οι ασυμφωνίες εδώ πέρα γιατί ξεχάστηκε από ό,τι φαίνεται σε κάποιες συνθήκες στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας. Αλλά ε, είναι πολιτικό το ζήτημα, γιατί το καθαρά νομικό ζήτημα ε, έχει κρυθεί από ό,τι φαίνεται. Αλλά το πολιτικό παραμένει ανοιχτό. Και η πρότασή μου είναι να το κρατήσουμε ανοιχτό, να κρατήσουμε ανοιχτή την αναφορά δηλαδή και να ζητήσουμε μια τοποθέτηση από την Επιτροπή Απασχόλησης. Γιατί είναι αρμόδιες επιτροπές και μπορούν να ασχοληθούν με την πολιτική πτυχή του ζητήματος. Καλώς, οι κανόνες λένε ότι εφόσον ε, ένας ευρωβουλευτής ζητάει να μείνει ανοιχτή μια αναφορά και μάλιστα εδώ όπως το ζητάει ο πιτεζιάρ μένει ανοιχτή αναφορά. Πάντως εσείς έχετε τον τελευταίο λόγο, οπότε αν θέλετε κάτι ακόμα να πείτε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή σε εμά, στον κύριο Γιάρ, παρακαλώ. Θα ήθελα να απαντήσω σε αυτό το οποίο είπε η σε εμα στον κυριο γιαρ παρακαλω θα ηθελα να απαντησω σε αυτο το οποιο ειπε η η Κομισιόν είπε πως υπήρξε απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου του ILO, του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας στη Γενέβη. Το θέμα είναι εδώ πέρα πως δεν είναι πάντα σαφές το εάν το διοικητικό δικαστήριο αυτό του ILO στη Γενέβη σε αντίθεση με το ΔΕΚ μπορεί να αποφασίσει για έναν κανόνα του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης ενός διεθνούς οργανισμού. Για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ήταν σαφές πως το Ευρωπαϊκό Πρώτο Δικαιοπροδοκείο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είχε την αρμοδιότητα να αποφασίσει για την ισχύ κανόνων ε, του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της ΕΚΤ. Δεν ξέρω εάν ε, γνωρίζετε την ε, απόφαση 2870 στην οποία αναφέρθηκε από τη φαίνεται Κομισιόν, εκεί πέρα αναφέρονταν πως το Ευρωπαϊκό Γραφείο Ευρεσιτεχνίας δεν ήταν σίγουρο ας πούμε για το εάν το διοικητικό δικαστήριο ήταν αρμόδιο για να αποφασίσει για την ισχύ ενός κανόνα του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασής μας. Νομίζω πως το δικαστήριο του ΑΕΛΟ της Γενέβης είναι κατά κύριο λόγο αρμόδιο να αποφασίσει για την ερμηνεία του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης ε, του Γραφείου Ευρεσιτεχνιών. Εάν λοιπόν αμφισβητείτε το πώς πρέπει να ερμηνευθεί ένας κανόνας, είναι σαφές πως το Διοικητικό Δικαστήριο της Γενέβης έχει αρμοδιότητα. Αλλά όταν το ζήτημα είναι το εάν ένας κανόνας που περιέχεται στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης, ο ίδιος ο κανόνας αυτός ε, είναι σύνομος ή αποδεκτός ας πούμε, τότε τουλάχιστον το Ευρωπαϊκό Γραφείο Ευρεσιτεχνίας το, το, η δικιά μου υπηρεσία, το δικό μου γραφείο μάλιστα, αμφισβήτησε την αρμοδιότητα ε, και είναι σε αυτή την απόφαση που ερθει να διαβάσει η Κομισιόν, αμφισβήτησε την ε, αρμοδιότητα του Διοικητικού Δικαστηρίου της Γενέβη για το εάν και κατά πόσο μπορεί να κρίνει την ομότητα των λόγων κανόνα. Και στο τέλο αυτής της απόφασης το Διοικητικό Δικαστήριο λέει καθώς πρέπει να απορριφθούν επί της ουσίας δεν χρειάζεται να κρίνουμε τον τύπο των επιχειρημάτων ε, του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Βεστέχνης. Κάτι το περίεργο γιατί θεωρεί το Ευρωπαϊκό Γραφείο Ευρεσιτεχνών πως το Διοικητικό Δικαστήριο δεν μπορεί να κρίνει. Μετά κρίνει το Διοικητικό Δικαστήριο, αλλά δεν κρίνει το παραδεκτό του αιτήματο και λένε «Α, δεν έχει πια σημασία». Και άρα εγώ συμπεραίνω πως πράγματι δεν είναι θέμα αυτού του Διοικητικού Δικαστηρίου να, να πάρει αυτή την απόφαση και Άρα το ζήτημα έπρεπε να παραπενθεί στο δουσού του Ευρωπαϊκού Γραφείου Ευρεσιτεχνιών. Στα κράτη-μέλη δηλαδή με άλλα λόγια. Ευχαριστώ. Όπως και να έχει το πράγμα, όπως είπαμε και πριν, η αναφορά παραμένει ανοιχτή. Γιατί το ζήτησε ο κύριος Γιάρ. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ. Ερχόμαστε στην αναφορά αριθμό 18, αναφορά 1031 του 2010 του Κριστόφμου Φιλικικής Σταγέννη σχετικά με τη διακριτική μεταχείριση σε βάρος των μη Γάλλων Ευρωπαίων Επικών, όπως προκύπτει από τα δίδακτρα που επιβάλλει ο Οργανισμός Γαλλικής εκπαίδευση στο εξωτερικό. Εδώ μου λένε ότι η Καρολίν Πανσάν που είναι μέλος ε, του Κοινοβουλίου των Βρυξελών είναι εδώ για να μας παρουσιάσει αυτή την αναφορά. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι Ευρωβουλευτέ, εγώ ε, αντιπροσωπεύω τον κύριο Μό που είναι Βέλγο υπήκο και κατοικεί στην, στον Νίγηρα. Θα είμαι αρκετά σύντομη, αλλά θα ήθελα να σα παρουσιάσω την κατάσταση τη εν λόγω αναφορά. Η υπηρεσία για τη γαλλική εκπαίδευση στο εξωτερικό παριθμεί πολλά εγκαταστάσει, 486 ε, λύκεια, γαλλικά λύκεια σε διάφορε χώρε του εξωτερικού και η πρόσβαση στα σχολεία αυτά ε, υπόκειται στην καταβολή πολύ διδάκτρων που διαφέρουν ανάλογα με την εθνικότητα, την υπηκότητα του μαθητή. Πάντως για τα σχολεία που είναι εγκατεστημένα εκτός ε, της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Ο κύριος Μούνς κατοικεί στην ΙΑΜΕ και τα παιδιά του για μια σχολική χρονιά στην ΙΑΜΕ το Γαλλικό Λύκειο ζητά από τους Γάλλους υπηκόους 2.900 ευρώ δίδακτρα ενώ για τους μη Γάλλους υπηκούς, δηλαδή Βέλγους και Λιπους, από άλλες ευρωπαϊκές εθνικότητες, αυτά τα δίδακτρα ανέρχονται στα 4.100 ευρώ. Ε, προφανώς λοιπόν κατά την άποψη του κυρίου Μούνς και κατά την άποψη άλλων κατοίκων μη Γάλλων σε άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης πρόκειται σαφώς για μια διάκριση που βασίζεται στην εθνικότητα, στην υπηκότητα και εγώ ως, Ευρω... βουλευτής στο, στο γαλλόφωνο ε, κοινοβούλιο της... των Βρυξελών ε, έχω επαφή και με άλλους Βέλγους υπηκόους και Έκτοτε από το 1997 έχω ασχοληθεί με το θέμα και έχω ενημερώσει τους υπουργούς ε, αρμόδιους για αυτά τα θέματα. Θα ήθελα να σας πω, λοιπόν ότι οι γαλλικές αρχές ισχυρίζονται απέναντι στους μη Γάλλους υπηκούς ότι αυτά τα σχολεία είναι σχολεία ε, ανεξάρτητα. θα θέλαμε μόνο να θυμίσουμε τις αποφάσεις του 10 για παράδειγμα την απόφαση Γραβιέ και τα λοιπά που αφορούσε τα δίδακτρα που ζητούσαν ε, οι ανώτατες σχολές και τα βελγικά πανεπιστήμια ήταν επίσης ανεξάρτητα ιδιωτικά πανεπιστήμια ιδρύματα, αλλά οι εθνικοί κανόνες ισχύουν και για αυτά τα ιδρύματα, δεν είναι δηλαδή ισχύουν αυτό το επιχείρημα. Έπειτα για τα γαλλικά λύκεια που είναι, βρίσκονται εγκαταστημένα σε, ε, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισχύουν τα ίδια δίδακτρα. Όταν η Γαλλία θέλει λοιπόν να εφαρμόσει αυτό το, το, το σύστημα, το εφαρμόζει. Και επίσης θα πρέπει να δούμε αν ε, τα <laughs> σχολικά ιδρύματα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να εφαρμόζουν τους ευρωπαϊκούς κανόνες ε, κατά των διακρίσεων. Ήδη υπήρξαν σχετικές αποφάσεις του ΔΕΚ, όπως η απόφαση Wallraff που, που συμπεράνει ότι η ισότητα μεταχείρισης και η μη διάκριση ισχύει και εκτός ε, της επικράτησης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έπειτα εγώ θα ήθελα και να πω Δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετική η απάντηση κατά τη γνώμη μου. Θα πρέπει λοιπόν αυτή η εθνική, η ευρωπαϊκή υπηκότητα και η η έλλειψη διακρίσεων να ισχύει και για αυτά τα γαλλικά ιδρύματα που είναι εγκαταστημένα εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να κλείσω λέγοντα απλά ότι το ξέρουμε ότι η κατάργηση των διακρίσεων και του δικαιώματος στην παιδεία επί τη βάση της ε, υπηκότητας επιφέρει κόστος για τα κράτη και για τα σχολικά αυτά ιδρύματα. Αλλά πιστεύω πως η κατάργηση των διακρίσεων ισότητα μεταχείρισης θα αξίζει τον κόπο να εφαρμόζονται οι ευρωπαϊκοί κανόνες στα σχολικά ιδρύματα που είναι εγκαταστημένα στο εξωτερικό από τη στιγμή που εξαρτώνται από ένα από τα κράτη-μέλη. Ε, πιστεύω πως η Επιτροπή σας είναι ένα πολύ ωραίο παράδειγμα άμεσης ε, δημοκρατίας. Θα μπορούσε να έχει στραφεί στο 10 ο κύριος Μούνς, αλλά πιστεύω πως ε, το πέρασμα από την Επιτροπή σας είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί βασίζεται στη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Κομισιόν για να μπορέσει να εξελιχθεί η, νομοθεσία της Γαλλικής Δημοκρατίας. Σας ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Κομισιόν. τον Βάλτε Σαβιέρη. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Όντως γνωρίζουμε αυτή την κατάσταση. Ε, πολύ ωραία την παρουσίασε η αναφέρουσα. Εμείς έχουμε αρχίσει εντατικό διάλογο με τις γαλλικές αρχές που επίσης θέλουν, είναι πρόθυμες για διάλογο μαζί μας. Έχουμε ανταλλάξει διάφορες επιστολές, έχουν υπάρξει ε, συνεδριάσεις, θα γίνουν και άλλες και σύντομα θα ληφθεί απόφαση μέχρι τις αρχές του επόμενου χρόνου, πιστεύω. Τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο περιμένουμε ότι θα ληφθεί απόφαση. Εγώ έχω μια ερώτηση. Γιατί παίρνει τόσο χρόνο. Να σας πω γιατί. Γιατί υπάρχει μια υποχρεωτική φάση στην φάση προ της ε, διαδικασίας κατά παράβαση. Είμαστε υποχρεωμένοι να ξεκινήσουμε διάλογο μέσω του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαλόγου για άτυπο διάλογο με το κράτος μέλος. Γιατί και χρειαζόμαστε και περισσότερες πληροφορίες. Γιατί όπως τόνισε η αναφέρουσα υπάρχει το θέμα του κατά πόσο ισχύει η συνθήκη μας εκτός της Ένωσης. Διότι ορισμένα από αυτά τα ιδρύματα είναι ας πούμε σε έμεση διαχείριση. Αν δεν ληφθεί απόφαση, έχουν υπάρξει αποφάσεις του ΔΕΚ όντως, αλλά μόνο από τη στιγμή που υπάρχει επαρκή σύνδεση ανάμεσα στην κατάσταση εκτός της Ένωσης και, μια, ε, και ένα σημείο εντός Ενώσεως. Δεν είναι προφανές δηλαδή ότι άμεσα ισχύει η συνθήκη. Αυτά συζητάμε με τις γαλλικές αρχές. Μάλιστα, κατάλαβα. Μάλιστα. Ο κύριος Γιάρα έχει ζητήσει το λόγο. Έχετε το λόγο. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, χοντρικά να τα πω. Εάν είναι, αν είναι σωστό αυτό το οποίο συμβαίνει, ξεχάσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ πέρα εντελώ που θέλουμε να δημιουργήσουμε και ευρωπαϊκή υπηκότητα κτλ. Και, και ξαφνικά έχουμε εδώ πέρα διακρίσεις σε άλλη χώρα. Δηλαδή πρέπει να αναλειτουργεί στο εσωτερικό το, το σύστημα. Πρέπει να υπάρχουν τα, τα βασικά δικαιώματα των, Ευρωπαίων πολιτών. Εγώ, αλλά εγώ δεν είμαι νομικός βεβαίως. Οι νομικοί βρίσκουν εκεί πέρα παραθυράκια, αλλά για μένα είναι ξεκάθαρη περίπτωση διακριτικής μεταχείρισης. Η Κομισιόν με την επικοινωνία, με το διάλογο που είχε τώρα με την Γαλλία, ακούω πως δεν είναι ικανοποιημένη και αναμένει πληροφορίες, οπότε πρέπει να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά αλλά θέλω να συμφωνήσω εδώ πέρα με τον πρόεδρο και να παρακαλέσω την Κομισιό να, να κινητοποιηθεί. Γιατί αλλιώ θα πρέπει να, να κινηθεί νομικά ο άνθρωπο. Ο Γιατί, τι γίνεται, Μες έχουμε διαφορετικά καθεστώτα εντό της Ευρωπαϊκή Ένωση λάμπει ο ήλιος και μετά εκτός ό,τι, ό,τι θέλουμε γίνεται. Εγώ σκέφτομαι δηλαδή, ήμουνα και μέχρι τώρα πούμε, αρκετά αφελή, ώστε σκεφτόμουν ότι αν βρεθώ σε μια τρίτη χώρα μπορώ να πάω σε μια γαλλική πρεσβεία και να πω, ξέρετε, εντάξει, μπορεί να είμαι Γερμανό, αλλά είμαι υπήκο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και να μου βοηθήσουν. Αλλά από ό,τι φαίνεται εδώ πέρα δεν ισχύουν τα, τα βασικά. Ναι. Όπω ξέρετε, Είπε ότι θέλει να μείνει ανοιχτή η αναφορά σας. Θα μείνει ανοιχτή. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι ακόμα. κλείνοντα. Ναι, πολύ σύντομα. Ευχαριστώ καταρχήν για τις παρεμβάσεις σας που είναι θετικές. Ελπίζω πως η Κομισιόν θα είναι αρκετά αυστηρή και θα πει ότι όντως η μη διάκριση θα πρέπει να επικρατήσει όσον αφορά την πρόσβαση στα λύκεια και στην παιδεία. Γιατί, εντάξει, χρειάζονται όρια, ε, χρειάζονται δεσμεύσεις. Όπως οι αποφάσεις του ΔΕΚ ήταν δεσμευτικές για τα βελγικά πανεπιστήμια, το ίδιο θα πρέπει να γίνει, γίνει και για αλλού. Πολλά παιδιά από αυτά κοντεύουν να φτάσουν στη σύνταξη από τότε που ασχολούμαι με το θέμα. Πρέπει πλέον να δουλέψει, να, να, να γίνει κάτι. Ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε στην επόμενη αναφορά που είναι η 358 του Νέρισον του Πορτοκαλικής Αγένειας σχετικά με τα ασφαλιστικά του δικαιώματα. Μου αναφέρον δεν είναι εδώ και γι' αυτό στρέφομαι στην Κομισιόν. Ο κύριος Μαυρίδη. Καλό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως ξέρετε, κατόπιν αυτής της αναφοράς η Κομισιόν ε, ξεκίνησε μια διαδικασία κατά παράβαση και το αποτέλεσμα ήταν ότι η Ολλανδική νομοθεσία άλλαξε. Από την 1η η 2012. Αντίθετα, η διαδικασία κατά παράβαση κατά των κάτω χωρών δεν κατέληξε γιατί το δικαστήριο απέρριψε την προσφυγή. Εν τω μεταξύ, δεύτερη μου παρατηρήση είναι ότι μέσα σε μία απόφαση του 10 στην υπόθεση Σαλμίνγκ, το δικαστήριο απεφάνθη ότι το, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισχύει για τους εργαζόμενους που εργάζονται στις πλατφόρμες εξόριξης που βρίσκονται στα ανοιχτά των κάτω χωρών. Είναι μια πολύ σημαντική απόφαση και μετά από αυτή την απόφαση του δικαστηρίου ε, χαιρετίζουμε το θάρρος των, του αναφέροντος που συνεχίζουν τη διαδικασία σύμφωνα με τις διαδικασίες και τις προθεσμίες που προβλέπονται από το Διεθνές Δίκαιο ενώπιον των αρχών της κάτω, των κάτω χωρών που είναι υποχρεωμένες να σέβονται το κοινοτικό δίκαιο όπως αυτό ερμηνεύεται από το ΔΕΚ στην υπόθεση Σαλεμίνγκ. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστούμε. Σχόλια. Αφού δεν υπάρχουν σχόλια, εντάξει, κλείνει. Και φτάνουμε στο σημείο 20. Αναφορά 76-2012 του Μάρκ Όστιν, Βρετανικής Ιθαγένειας. Μου λένε ότι δεν είναι παρόν ο αναφέρον. Θα δώσουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο αναφέρον δεν είναι εδώ. Θα σας παρουσιάσω εγώ κάπως ε, σύντομα το θέμα. Ο αναφέρον, λοιπόν, αγοράζει πολιτιστικά αγαθά, αντίκες ή τέλος πάντων ε, παλιά αντικείμενα στο χώρο, στη χώρα μέλος που ονομάζει Β και στην Έχεια εισάγει στη χώρα μέλος Α όπου κατοικεί από ό,τι φαίνεται τα αντικείμενα αυτά και εκεί στη χώρα Α προσφέρει τα αγαθά αυτά σε άλλους καταναλωτές μέσω ενός ε, μιας ιστοσελίδας τύπου eBay. Ποιο είναι το πρόβλημα τώρα ότι ο αναφέρον λέει πως για κάθε έργο τέχνης το κράτος μέλος Α απαιτεί άδεια για να μπορέσει να εξάγει τα εν λόγω αγαθά. Από τη μια πρέπει να πούμε ότι ο αναφέρον λέει πως τα εν λόγω αγαθά δεν έχουν καμία ιστορική αξία για τη χώρα μέλος Α και ότι πρόκειται για αγαθά μιας ε, χαμηλής αξίας αντικείμενα. Επίσης, Πρέπει να παρατηρήσουμε εδώ ότι ο αναφέρον υποστηρίζει επίσης πως ε, άλλοι οικονομικοί φορείς που είναι ανταγωνιστές του γραπτά έχουν πει και έχουν δημοσιεύσει πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες δεν απαιτείται τέτοια άδεια. Οπότε τελικά δεν ξέρουμε πολύ καλά ποια ακριβώς είναι η κατάσταση σε αυτή τη χώρα μέλος Α και αγνούμε πλήρως και την ταυτότητα της ενδιαφερόμενης χώρας. Στα πλαίσια αυτά, ο αναφέρον ζητάει νομική γνωμοδότηση για αυτό το οποίο ο ίδιος παρουσιάζει ως σενάριο. μια υποθετική κατάσταση. Όσον αφορά το ευρωπαϊκό δίκαιο, η κατάσταση πάντως είναι αρκετά σαφής, διότι τα αντικείμενα ε, αυτά οι αντίκες δεν εναρμονίζονται, δεν τυχαίνουν ε, μεταχείριση σύμφωνα με το παράγωγο δίκαιο και είναι κάτι που έχει να κάνει με τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή τα αντικείμενα 35, τα άρθρα 35 και 36 της συνθήκης διέπουν την κατάσταση αυτή. Το άρθρο 35 απαγορεύει τον ποσοτικό περιορισμό ή αντίστοιχες ε, απαγορεύσεις στην εξαγωγή. Το άρθρο 36 προβλέπει περιορισμούς και κάποιες εξαιρέσεις στο άρθρο 35 εάν το κράτος μέλος μπορεί να τα αιτιολογήσει. Η αιτιολόγηση που μας ενδιαφέρει εδώ πέρα είναι η προστασία των εθνικών θησαυρών που έχουν μια καλλιτεχνική, ιστορική ή αρχαιολογική αξία. Η απάντηση δηλαδή θα ήταν ότι σε γενικό κανόνα η, τα καθεστώτα διαδότησης, οι διάφορες διατυπώσεις είναι κάτι δυνατό βάσει της ηθίκης, αλλά πρέπει να πούμε πως κάθε κράτος μέλος καθορίζει από μόνο του τι θεωρεί εθνικό θησαυρό. Κάθε χώρα μέλος δηλαδή πρέπει να πει ποια είναι τα αγαθά τα οποία ανταποκρίνονται ε, στον όρο αυτό. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο πάντως μέχρι τώρα δεν είχε την ευκαιρία να αποφανθεί επί του όρου αυτού εθνικός θησαυρό, ο οποίος συνεπώς επιδέχεται ε, διάφορες ερμηνείες. Και άρα είναι πολύ δύσκολο να απαντήσουμε με περισσότερες λεπτομέρειες στην ερώτηση του αναφέροντος, εφόσον δεν μας εξηγήσει πιο συγκεκριμένα τις πραγματικές συνθήκες που ισχύουν στη χώρα μέλος Α και εφόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ξέρει τελικά ποια είναι αυτή η χώρα. Σας ευχαριστώ. Eh, Ευχαριστούμε. Σχόλια, παρεμβάσεις. Οπότε σε αυτή την περίπτωση εγώ θα έλεγα ότι μια που δεν είναι και παρόν ο αναφέρον να στείλουμε κάτι στις αρχές της Πορτογαλίας και ανάλογα με την απάντησή τους να ολοκληρώσουμε την εξέταση της αναφοράς αυτής. Και περνάμε στο σημείο 21. Αναφορά 1386 του 2011 του Αντώνιο Χαβιέ Ροντρίγκε Καστίγιο. Η Ισπανική Σταγέννη σχετικά με το καθεστώ υποχρεωτικών διοδίων στον αυτοκινητόδρομο Via do Infante στην περιοχή του Αλγκάρβε τη Πορτογαλία. Εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο κύριο Ράσμουσεν έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε ο αναφέρον, όπως αναφέρει, είναι αντίθετος με τα υποχρεωτικά διόδια που έχει επιβάλει η πορτογαλική κυβέρνηση σε αυτοκινητόδρομο στο Αλγάρβε. Η απάντηση της Κομισιόν είναι απλή και σύντομη. Τα διόδια στους αυτοκινητόδρομους είναι ζήτημα οδηγίας ε, 1999 κάθετο 62 κάθετο Ευρωπαϊκή Κοινότητα και αφορούν φορτηγά Η Κομισιόν έχει λάβει λοιπόν πολλές καταγγελίες και έχει ξεκινήσει η διαδικασία επί παραβάση κατά της Πορτογαλίας ε, η οποία ακόμα δεν έχει εκδικαστεί και άρα η Κομισιόν δεν έχει ε, ακόμα καταλήξει κάπου. Ε, εν πάση να αναμένεται σύντομα απόφαση, οπότε δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της διαδικασίας. Όσον αφορά τα επιβατικά γεωταχή, που επίσης αναφέρονται στην επιστολή του αναφέροντος. Δεν υπάρχει νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πέρα από τις γενικές αρχές της συνθήκης ε, που αναφέρουν πως δεν μπορεί να υπάρξει διακριτική μεταχείριση για μη κατοίκους. Εκεί η Κομισιόν έχει κάνει τις ερευνές της και δεν έχει βρει κάποιο λόγο ε, για να κινηθεί κατά της Πορτογαλίας. Σας ευχαριστώ. Ε, Αντιλαμβάνομαι τις ανησυχίες σας για την κατάσταση διοδίων ανάμεσα στην Ισπανία και την Πορτογαλία ενώ υπήρχε η ελευθερία διακίνησης έτσι κι αλλιώς όμως στην Επιτροπή εκρεμεί ακόμα το θέμα, άρα μένει ανοιχτή η αναφορά μέχρι να λυθεί το θέμα αυτό της τοποθέτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρος. Λοιπόν, τώρα έχουμε την ε, αναφορά 923-2011 από λιθουανική ηθαγένεια αναφέρουσα σε σχέση με την οδηγια 2038. Η αναφέρουσα δεν είναι παρούσα, οπότε θα δώσω το λόγο στην Κομισιόν για να μας δώσει τη θέση της. Η Καρολίν Λουπ. Σας ευχαριστώ. Η αναφέρουσα είναι λιθωνικής ηθαγένειας ε, και κατοικεί στο Γιβραλτάρα θέλει η σύζυγος είναι ουκρανικής ηθαγένειας και ήθελε να επιστρέψει στην, ε, να επισκεφτεί τη χώρα της. Ζήτησε μια θεώρηση η οποία δεν της δόθηκε. Μια τέτοια απέτηση θεώρησης είναι αντίθετη από το, με το άρθρο 2 παράγραφος 6 ε, της οδηγιας 2004 2004-38 και κατά τη γνώμη στην απάντησή μας αναφέραμε ότι περιμέναμε τροποποίηση στην σχετική νομοθεσία της Λιθουανίας που έπρεπε να εφαρμόσει την σχετική νομοθεσία από τις 29 Απριλίου του 2004. Λάβαμε την τροποποίηση στις 30 Ιουνίου 2010 και κοινοποιήθηκε στην Κομισιόν στις 27 Ιουλίου και τώρα η νομοθεσία είναι πλέον ξεκάθαρη. δεν είναι υπήκος κράτος μέλους, αλλά είναι, έχει στην κατοχή του κάρτα παραμονής ενός κράτους της Ένωσης μπορεί να παραμείνει χωρίς θεώρηση στα κράτη-μέλη της ε, Ένωσης για τρεις μήνες. Αν ο θέλει να επιστρέψει λοιπόν στη Λιθουανία για επίσκεψη, η σύζυγός του δεν χρειάζεται να έχει θεώρηση πλέον. Άρα λοιπόν, επί τη βάση αυτών των πληροφοριών της Κομισιόν, καταλήγουμε ότι έχει λυθεί το θέμα. Έχει ξεπεραστεί το πρόβλημα. Α, θα πρέπει να ενημερώσουμε για αυτές τις πληροφορίες που πήραμε από την ε, Κομισιόν και να επαληθεύσουμε τι έγινε μετά στην πράξη, αν όντω η κατάσταση έχει αλλάξει ή όχι. Πιστεύω ωστόσο ότι επί τη βάση αυτών των πληροφοριών που δεν είναι ε, πλήρης, είναι καλό να αφήσουμε ανοιχτή την αναφορά αυτή και να προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε περαιτέρω για να δούμε και ο, ο αναφέρον τελικά τι έκανε. Δεν υπάρχουν ε, άλλα σημεία στην ημερήσια διαταξή. Μόνο αν υπάρχουν ε, ανακοινώσει για το δεύτερο τμήμα, το τμήμα Β. Υπάρχουν. Έχουμε κάποια ανακοίνωση στο τμήμα Β, την υπαρθμό 33, από πλευράς του συναδέλφου Τζανόκα, που και μεταφέρεται στο τμήμα Α. Σας ευχαριστώ, δεν έχουμε άλλα σημεία στη διάταξη, οπότε κλείνει αυτή η συνεδρίαση.